M. Poussek est dans le taxi de l'aéroport. Il arrive à chaque moment. Bene. Cominciamo. Καλημέρα σας, να ξεκινήσουμε. Και επειδή το πρωινό είναι πλούσιο, Βλέπετε και τις καμπίνες και οι γλώσσες φαίνονται στα τζάμια από τις καμπίνες. Qual è il numero della, per la Lituania? Perché peut le dire parce non je ne le Bene. Benvenuti να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη σημαντική κοινή συνεδρίαση. Από ό,τι βλέπω δεν έχετε βρει ακόμη τα κανάλια για τη διερμηνία. mais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 είναι το κανάλι για τηλεφωνικά. Allora, benvenuti a tutti i partecipanti. Καλώς ορίσατε σε αυτή τη σημαντική κοινή συνεδρίαση που συνδιοργανώνεται από την Επιτροπή Βιομηχανίας και την Προεδρία, τη Λιθωνική Προεδρία του Συμβουλίου. Θα ήθελα ιδίω να καλωσορίσω τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που ήρθαν στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσουν τη συνάντηση αυτή και θα πάρουν το λόγο κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας ε, για να συνεισφέρουν στη συζήτηση. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδίως την Προεδρία της Λιθουανίας και τον Πρόεδρο Ζεμαϊτάιτης που πρότεινε την πρωτοβουλία αυτή. Πρόκειται για ένα ζωτικό θέμα για το παρόν και για τον μέλλον μας. Πρόκειται για την εσωτερική αγορά ενέργειας. Τέτοιες πρωτοβουλίες που οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και της Εκπεριτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου αποτελούν σημαντική έκφραση της διαθεσμικής και διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή συνεδρίαση δίνει μια εξαίρετη ευκαιρία για την ανταλλαγή ειλικρινών και σβάθος απόψεων μεταξύ των εθνικών βουλευτών και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ενεργειακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ζωτική του σημασία. Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πράγματι σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας είναι απόλυτη προτεραιότητα και σε ό,τι αφορά την υποδομή, αλλά και σε ό,τι αφορά την, το μεγαλύτερο ανταγωνισμό και την πτώση των τιμών. Υπάρχουν όμως καθυστερήσεις σε όλες τις χώρες, σημαντικές διαφορές ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων, πάρα πολλές διαδικασίες, κατά παραβάση διαδικασίες ακόμη και μια οικονομική συγκυρία η οποία απαιτεί άμεσες λύσεις που να δώσουν και μακροπρόθεσμες προοπτικές. Σίγουρα η συζήτηση θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική. Η την πρωινή συνεδρίαση θα την προεδρεύσω εγώ και ο κύριος Ζαμαϊτάιτης ε, θα συντονίσει την απογευματινή συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 3 το απόγευμα. Το λόγο θα δώσω τώρα στον κύριο Ζαμαϊτάτης, ε, ο οποίος ε, είναι πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του ΣΕΜΑΣ της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, προσκεκλημένοι, κύριε και κύριοι, η οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα είναι οι μεγάλοι στόχοι της Ένωση και πολύ σημαντική σήμερα, όπου ολόκληρη η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η βιώσιμη ενέργεια και οι όχι υψηλέ τιμέ είναι βασική στόχη επίση. Το Φεβρουάριο του 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε και πάλι τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής, δηλαδή ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας και διασφάλιση ότι μετά το 2015 δεν θα αντιμετωπίσουμε, ή μάλλον δεν θα έχουμε πλέον νησίδες απομονωμένες ενέργειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει γίνει, το Μάιο φέτος το Συμβούλιο χρειάστηκε να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή των στόχων μέχρι τέλος του έτους αποφάσισε δηλαδή, και να δώσει επισκόπηση της ενεργειακής πολιτικής, να διασφαλίσει ισότιμους όρους για τους παραγωγούς ενέργειας. Τονίζω ότι η βιωσιμότητα της παραγωγής ενέργειας και η ολοκλήρωση των, ε, η ενοποίηση μάλλον των συστημάτων παραγωγής ενέργειας για την δημιουργία της ενιαίας αγοράς και για να διασφαλιστεί και η εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής. Αυτή είναι η βασική στόχη της Λιθουανικής Προεδρίας και σημειώνω με ικανοποίηση ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας εγκρίθηκαν δύο σημαντικότατες εκθέσεις. Αφενός η έκθεση που επιγράφεται πρόοδος στην ολοκλήρωση της εννέας αγοράς ενέργειας και επίσης ή αλλαγέ που θα επιφέρει στην εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής. Θέλω να τονίσω ότι τα έγγραφα αυτά εγκρίθηκαν για πρώτη φορά παρόμοια έγγραφα, δηλαδή στο Συμβούλιο Υπουργών. Η Λιθουανία κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες στη διάρκεια της Προεδρίας της, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την ε, πορεία προς την ενιαία αγορά και την διάσταση της εξωτερικής πολιτικής. Και είμαι βέβαιος ότι τα κείμενα αυτά θα αποδειχθούν σημαντικά και για το μέλλον όταν θα κληθούμε να λάβουμε και άλλες αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα αγαπητές και αγαπητοί να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Πρόεδρο κυρία Σαρτόρη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε, για την συνεισφορά της και τις προσπάθειες που κατέβαλε για την διοργάνωση της σημερινής πολύ σημαντικής κοινή συνεδρίασης. Θα ευχαριστήσω την κυρία Σαρτόρη και για την προσωπική της δέσμευση και εμπλοκή και στην πρόσκληση ιδιαίτερα των εθνικών βουλευτών για να συζητήσουν πολύ σημαντικούς ενεργειακούς στόχους. Απευθύνω λοιπόν και πάλι ένα θερμό καλώς ορίσατε σε όλες και όλους εσάς και εύχομαι και σε εσάς και σε εμάς καλή επιτυχία στις εργασίες μας. Ευχαριστώ. Βερμά τον συνάδελφο, τον κύριο Σεμαϊκάτης, για την ε, παρουσία του εδώ και για το χαιρετισμό που μας απίφθηνε. Και προφανώς υπάρχουν ε, και μέλη από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την παρουσία τους εδώ και χαιρετίζω και όλα τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τώρα, να περάσουμε στις παρεμβάσεις. θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 11 και 20, προκειμένου να έχουμε και τη δυνατότητα συζήτησης. Επομένως, θα ξεκινήσουμε τώρα με μια παρέμβαση 10-15 λεπτών. και θα ήθελα να σας ζητήσω να μιλάτε και αργά για να διευκολύνετε τους διερμηνείς. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιάροσλαφ Νεβέροβιτς, τον Υπουργό Ενέργειας της Συμφωνίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού εξότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την δυνατότητα που μου δίνετε να παρευρεθώ εδώ μαζί σας και να συζητήσουμε την ε, πρόοδο που επιτυχαίνουμε προς την ολοκλήρωση της ε, αγοράς ενέργειας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το θέμα. Και εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ε, ιδέες και προτάσεις από πλευράς Συμβουλίου σε ό,τι φορά την ενεργειακή πολιτική. Ουσιαστικά το θέμα είναι πώς ακριβώς θα έχουμε αυτή την ενιαία εσωτερική ενεργειακή αγορά με την ενσωμάτωση 28 διαφορετικών εθνικών αγορών σε μία. Θα ήθελα συντομία να επαναλάβω τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργικής Πολιτικής, που είναι η θέσπιση ενός βιώσιμου ενεργειακού ευρωπαϊκού συστήματος, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ε, ε, προσφοράς ε, στους πολίτες αλλά και στη βιομηχανία. Μια ανταγωνιστική λοιπόν, ε, αλλά και πλήρω ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά. Είναι μια κυρίαρχη προτεραιότητα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ε, να εξετάσουμε το θέμα τη ενεργειακή πολιτική. Τον Φεβρουάριο του 2011 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν ξεκάθαρα να ολοκληρωθεί η ενεργειακή αγορά μέχρι τα τέλη του επόμενου έτου και να απαλείψουν οποιοδήποτε τέτοιε νησίδε μετά το 2015. Κατά τη διάρκεια του Μαΐου, τη Συνόδου Κορυφή το Μάιο, το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να ε, καταγράψει τα στοιχεία που θεωρεί σημαντικά για την ε, επίτευξη των στόχων. Δεδομένη τη ε, αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών αγορών ενέργεια, κληθήκαμε να αναθεωρήσουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2011 για την εξωτερική διάσταση τη ενεργειακή πολιτική. Η Λιθουανική Προεδρία ανέλαβε ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και θέλησε να έχει και τις ε, παρεμβάσεις κομισιών και κρατών μελών. Χαιρόμαστε που το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση του κυρίου Βούζεκ για την ενεργειακή αγορά στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Κατόπιν των προσπαθειών μας ε, για την ολοκλήρωση της ενεργικής αγοράς και την ενίσχυση της εξωτερικής διάσταση τη ε, πολιτική μας, έχουμε δύο εκθέσεις ε, του Συμβουλίου που προετοιμάστηκαν και υιοθετήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τους Υπουργού Ενεργείας. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία, να τα εξετάζουμε και σε εθνικό επίπεδο, καθώ ε, προσπαθούμε να ε, επιτύχουμε του στόχου μα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτέ οι εκθέσει λοιπόν καταγράφουν το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και εντοπίζουν πού πρέπει να εστιάσουμε τι προσπαθίε μα ε, στο μέλλον. Εναρμόνιση κανόνων για την αγορά μαζί με άλλε υποδομέ για την ενέργεια. Αυτά αποτελούν τη βάση μια ολοκληρωμένη αγορά ενέργεια. Και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μπορώ να πω ότι ήδη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση τη αγορά, Ωστόσο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον τελικό μας προορισμό. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ τα, στα όσα υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέλη στην ε, έκθεση του Συμβουλίου. Χρειαζόμαστε περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς με πλήρη μεταφορά και εφαρμογή του τρίτου πακέτου ενέργειας μαζί με υιοθέτηση και εφαρμογή των ε, ε, κωδίκων δικτύου. Αυτό θα διασφαλίσει ένα συνεκτικό και σταθερό και βιώσιμο ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι ακρογωνίας λήθος μια ενοποιημένης αγοράς ενέργειας με ανταγωνισμό και ενεργούς πολίτες και καταναλωτές. Θα ήθελα εδώ να τονίσω τον ε, ρόλο αυτών των network codes που βασίζεται ακριβώς στην ρυθμιστική σύγκληση, την εναρμόνιση των κανόνων για ολόκληρο τον κλάδο. Αυτά τα στοιχεία είναι κρίσιμη σημασία για την διασφάλιση των ροών ενέργειας. Άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ανάπτυξη της ενεργειακής υποδομής, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά τέτοια ενιαία αλληλένδετη αγορά ε, για να παράσχουμε τις απαραίτητες ροές ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, επενδυτικές προκλήσεις, να συνδέσουμε τις ενεργειακές νησίδες και να ε, αποκαταστήσουμε τις καθυστερήσεις όπου αυτές υπάρχουν. Αυτό συνδέεται και με την εφαρμογή προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Τον Οκτώβριο η Κομισιόν υιοθέτησε το σχετικό κατάλογο και έχει ήδη παρουσιαστεί στο Βίλνιους στην ε, διάσκεψη ενεργειακής υποδομής στις αρχές Νοεμβρίου. Αυτή η διάσκεψη υψηλού επίπεδου ε, μας επέτρεψε να δείξουμε ακριβώς τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα ως Ευρώπη, ποιες προκλήσεις παραμένουν και ποιες λύσεις ε, μπορούν να βρεθούν για να ολοκληρώσουμε την ενεργειακή αγορά. Η κατάλληλη χρηματοδότηση και η περιφερειακή συνεργασία είναι κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχή εφαρμογή των PCIs αλλά και η αποδοχή από την κοινή γνώμη είναι σημαντικό θέμα και η διάσκεψη αυτή καθ' αυτή αξιοποιήθηκε για να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό για τα ευρωπαϊκά προγράμματα υποδομής. Η διαδικασία υιοθέτηση του καταλόγου PCI ελπίζουμε να ολοκληρωθεί μέχρι τον ε, Δεκέμβριο, μέχρι τα τέλη του έτους δηλαδή. Η υιοθέτηση του καταλόγου PCI σημαίνει ότι περνάμε στην φάση υλοποίηση των προγραμμάτων που είναι τόσο σημαντικά για την ιστορική αγορά και την ε, ολοκλήρωση των αγορών. Οι 248 PCIs ε, επιλέγησαν από 12 περιφερειακές ομάδες και άλλα περιφερειακά προγράμματα ε, για να διασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή διασύνδεση, διασύνδεση μεταξύ κρατών μελών. Έτσι, επιλύουμε σημεία συμφόρηση και στενώσεις για την ολοκλήρωση αγορά και πάνω από 5 δις θα ε, αφιερωθούν σε αυτό το σκοπό. χωρί την οικονομική αυτή στήριξη, τα προγράμματα υποδομών δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Και τα PCIs όταν υλοποιηθούν σίγουρα θα ε, συμβάλλουν στην απάλληψη των ενεργειακών συνείδων, της απομόνωσης ενεργειακής και τη διαφοροποίησης. Ε, στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις ε, πηγές ενέργειας και τους παρόχους. Ε, αυτό θα μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση και θα αυξήσει την ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διασφαλιστεί επίσης σε βαριά επίπεδο διασυνοριακής διασύνδεσης όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν το στόχο του 10% ε, στην ηλεκτρική ενέργεια. Στο φυσικό αέριο θα έχουμε επίσης σημαντικές αλλαγές. Νίμιον 1 είναι το πρότυπο ε, που θα υλοποιηθεί από την πλειονότητα των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε νέες ενεργειακούς πόρους, όλα τα κρατημέλη θα έχουν πρόσβαση τουλάχιστον σε δύο πηγές παρόχων. Τα PCI είναι απαραίτητα και από πλευράς περιεχομένου πέρα της μορφής. για την επίτευξη ενός επίπεδου διασύνδεσης και ο κατάλληλο του PCI ε, ενσωματώνει όλα αυτά τα συστήματα. Και εδώ αναφέρομαι ε, στο project που αφορά τις χώρες της Βαλτικής. Η εφαρμογή αυτού του project ε, θα διασφαλίσει ότι τα κράτη της Βαλτικής θα, θα ενοποιηθούν και θα συμμετάσχουν 100% σε αυτή τη νέα πολιτική. Έχουμε πλέον ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα με τα PCIs, ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα αλληλεγγύης και διασύνδεσης των περιφερειακών αγορών που θα ε, μας ενοποιήσουν περαιτέρω σε μία και μόνο εσωτερική αγορά. Είναι πολύ ξεκάθαρο το καθήκον μπροστά μας, η υλοποίηση αυτών των project προτεραιότητας. Χρειαζόμαστε επιτυχή συνεργασία και συμφωνία επιπρακτικών ρυθμιστικών ζητημάτων. Αυτές οι προκλήσεις πρέπει να επιληθούν πριν θεωρήσουμε ολοκληρωμένο το, το στόχο ε, της ολοκλήρωσης αγοράς. Όλα αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα προηγουμένως με τα network codes και ε, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των καταναλωτών. Είμαι σίγουρος ότι μέχρι το αίτιο του 2014 θα έχουμε ε, κάνει αποφασιστικά βήματα προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος αυτή με μονομερείς κινήσεις μπορούν να κατακαιρματίσουν την αγορά μας. Πρέπει να αποφύγουμε, να αποτρέψουμε ε, τέτοιες στευρώσεις, αν και κάποιες φορές ε, υπάρχουν και εθνικά μέτρα, όπως είναι η ε, επιδοτήσεις και μάλιστα υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ μας για αυτές τις επιδοτήσεις. Έτσι εμείς οι ίδιοι μπορούμε να βλάψουμε την εσωτερική αγορά με τον κατακαιρματισμό και τις τεντώσεις. Εδώ βλέπουμε θετικέ εξελίξει παρόλα αυτά. Πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν για, το, τη δημόσια παρέμβαση της ε, αγορές ενέργεια. Παρέχει ε, κατευθύνσει για τα νέα προγράμματα επιδότηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στις αγορές ενέργειας. Σε ό,τι φορά την επάρκεια παραγωγής ενέργειας, είμαι σίγουρος ότι και με, την, ε, ε, με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν αυτό θα γίνεται με έναν οικονομικά βιώσιμο τρόπο και χωρίς να θέτει, τίθεται σε κίνδυνο η αγορά της ενέργειας μια πιο πρωτότυπη προσέγγιση θα πρέπει να έχουμε και προ την αγορά τη ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ αναφέρομαι και στα κριτήρια τη εξάντα αναθεώρηση των όρων θέσπιση, μηχανισμού αποζημίωση για την ικανότητα. Ε, προσεκτική αξιολόγηση των κριτηρίων θα πρέπει να αποτρέψει στρεβλώσεις και ανεπάρκειε αγορά. Ε, μεγαλύτερη ανταπόκριση από πλευρά τη ζήτηση και ευελιξία. Πολύ σημαντικά στοιχεία για το μέλλον τη αγορά. Ε, η πλευρά της ζήτησης δηλαδή, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα μας επιτρέψουν ε, την... Ε, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και συμμετοχής στην αγορά για να επιτρέψουμε και τη βελτιστοποίηση των υποδομών και να αποφύγουμε δαπανηρές επενδύσεις. Έτσι προσδίδουμε περαιτέρω ευελιξία και αξιοπιστία ε, στο σύστημά μας. Ήδη έχουμε ένα καλό υπόβαθρο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα υποδομή ε, και ρυθμίσεων. Όλα αυτά μας θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να μεταφράσουμε τις προσδοκίες μας στην πραγματικότητα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ τον Υπουργό ενέργεια, τον κύριο Νεβέροβιτ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπούζεκ ο οποίος ε, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος ε, θα μιλήσει για το πώς ε, θα καταστεί λειτουργική η αγορά ενέργειας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί και αγαπητές φίλοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό που έχουμε μπροστά μας. Θέλουμε να μιλήσουμε για την ενέργεια που είναι τόσο σημαντική για τις οικονομίες μας και κυρίως επειδή θέλουμε να εκβιομηχανίσουμε ξανά την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, κάτι που φαίνεται να γίνεται απαραίτητο αν θέλουμε να κερδίσουμε σε ανταγωνιστικότητα σε όλο τον πλανήτη. Είναι λοιπόν τότε απαραίτητο να βελτιώσουμε την παραγωγή μας, μιλώντας γενικά. Και οι τιμές ενέργειας από την άποψη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικές. Υποστηρίζω απολύτως όλα όσα λέχθηκαν από τον κύριο Υπουργό που εκπροσωπεί την ε, Λιθουανική Προεδρία που φτάνει στο τέλος της αγαπητέ φίλε βεβαίως η Προεδρία σας αλλά έκανε πολλά πράγματα στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ενέργειας και επίσης σε μια προσπάθεια να κλείσει τα κενά μεταξύ των χωρών μελών και να προχωρήσει προς περισσότερες επενδύσεις υποδομών. Έχουμε λοιπόν κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Μετά από ένα εξάμεινο ε, μόλις ε, Λιθουανικής Προεδρίας βέβαια είναι και όλα τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρέπει να τονιστούν από την αρχή δηλαδή της θητείας της το 2009-2010 διότι ο διορισμός της Κομισιόν ε, άρχισε το 2010 και από τότε έγινε πολλή δουλειά νομοθετική προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας. Θα ρωτήσετε για ποιο λόγο. Θέλουμε να έχουμε διέξοδο, στρατηγή εξόδου από την κρίση. Δεν αρκεί η ανάκαμψη. Η σταθερότητα των ε, χρηματοπιστωτικών συστημάτων δεν αρκεί επίσης. Στρατηγική εξόδου σημαίνει ανάπτυξη έψιν 3 συν 4. Τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας γι' αυτό. Έχουμε την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρούμε σε μια ανανέωσή της με ξεπέρασμα 150 σημείων εχμής. Δεύτερο, καινοτομία, εκ νέου βιομηχανοποίηση της Ευρώπης με καινοτόμο οικονομία και βέβαια η ενέργεια. Η ασφάλεια προμήθειας ενέργειας, πολύ σημαντική αυτή, πολύ σημαντικό θέμα, φθηνές τιμές, δηλαδή ως το δυνατόν χαμηλότερες και βέβαια και προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να ληφθεί υπόψη. Επιτρέψτε μου να πω λοιπόν ότι η χρήση της εσωτερικής ή αγοράς ενέργειας της Ένωσης μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε και τα τρία στοιχεία. Πρώτα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλους τους ηθαγενείς πόρους, τους ε, ε, εσωτερικούς πόρους των χωρών μελών και να ανταγωνιστούμε στην ανοιχτή αγορά ενέργειας σε μια προσπάθεια να επιτύχουμε τις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Ταυτόχρονα πρέπει να συντονίσουμε την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι πολύ πιο ισχυρή η θέση μας στις διαπραγματεύσεις με τους εξωτερικούς προμηθευτές μας. ταυτόχρονα να φροντίσουμε να υπάρξει σταθερότητα των κανόνων στη μεγάλη αυτή αγορά ενέργειας της Ευρώπης. Ασφάλεια δικαίου δηλαδή, αλλά και βεβαιότητα ότι οι τιμές θα παραμείνουν στα επίπεδα που είναι. Για να οργανώσουμε την εσωτερική μας αγορά πρέπει να προσφέρουμε σταθερότητα τιμών στους επενδυτές. Εφόσον ενδιαφέρονται να επενδύσουν θα θέλουν να είναι βέβαιοι, λίγο πολύ τέλος πάντων, λίγο πολύ για την σταθερότητα των κανόνων και για τις μελλοντικέ τιμές ενέργειας. Δεν μπορεί αλλιώς να συντάξει κανείς επιχειρηματικό σχέδιο για μεγάλες επενδύσεις χωρίς τα στοιχεία αυτά. Θα πρέπει έτσι να οργανωθούμε λοιπόν στην ενιαία μας εσωτερική αγορά ενέργειας για να συμβάλλουμε να υπάρξει ασφάλεια, φθηνές τιμές, ανταγωνιστικές τιμές και βέβαια και προστασία περιβάλλοντος. Τι, ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η αγορά μας. Λίγα στοιχεία που φαίνονται να είναι τα πιο σημαντικά από την σκοπιά της έκθεσής μου, γιατί εγώ είμαι εισηγητής για την ενιαία αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από την έκθεσή μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτους δημοσίευσε ανακοίνωση με επιγραφή εσωτερική αγορά ενέργειας. Και η δική μου έκθεση αποτελεί την απάντηση στην ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι λοιπόν είναι απαραίτητο. Βεβαίως υποδομή, διαμεθοριακές διασυνδέσεις. Σεις κύριε Υπουργέ πριν από λίγα λεπτά δώσατε γενικά στοιχεία για το θέμα αυτό που αποτελεί μάλιστα και προτεραιότητα της Λιθουανικής Προεδρίας μέσα στην προτεραιότητα της ενέργειας. Πολύ σημαντική προτεραιότητα κύριε Υπουργέ, διότι χωρίς τις διασυνδέσεις αυτές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ενιαία αγορά ενέργειας. Χρειαζόμαστε αγωγούς, χρειαζόμαστε ηλεκτρικά δίκτυα, τα δηλαδή δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, που να διαβαίνουν τα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης. Έχουμε κάποια χρήματα. Έχουμε την ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη που ε, προβλέπει περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους αυτούς, τα χρήματα αυτά, για να δημιουργήσουμε τις πιο σημαντικές συνδέσεις. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους προς και προς Νότον γειτονές μας, σε μια ενεργειακή κοινότητα. Εννέα χώρες εν το σύνολο τρεις από την ανατολική γειτονία, δηλαδή Ουκρανία, Μολδαβία και Γεωργία και έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που δεν αποτελούν, τουλάχιστον ακόμη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταθέσουμε όλες τις προτάσεις μας και να ενωθούμε με τις δικές τους αγορές ενέργειας. Αυτό θα είναι πολύ θετικό και υπέρ της δικής μας ε, σταθερότητας για την προμήθεια της ενέργειας και για τη δική τους. Για την μεταφορά, για τους πόρους ενέργειας είναι πολύ σημαντικό να διευρυνθεί έτσι η αγορά μας και να χρησιμοποιηθούν σωστά και τα εθνικά μας χρήματα και τα χρήματα του ιδιωτικού τομέα σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις βεβαίως και η ευρωπαϊκή πόρη όπως είπα με την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Δεύτερο, χρειαζόμαστε κοινού κανόνες στην εσωτερική αγορά ενέργειας και πρώτον έντιμη, δίκαιη πρόσβαση στα δίκτυα, στους αγωγούς όλοι οι προμηθευτές ή αυτοί που φροντίζουν για την μεταφορά της ενέργειας να έχουν δίκαιη πρόσβαση, ε, έντιμη πρόσβαση στα δίκτυα αυτά. Είναι επίσης απαραίτητο αλλοδαπές εταιρείε από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν ε, που ε, θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας πρέπει να τους δώσουμε ασφάλεια ότι οι εσωτερικοί μας κανόνες είναι δίκαιοι και για αυτές. Χρειαζόμαστε κώδικες για τη μεταφορά και διανομή που να είναι συγκρίσιμοι. Γιατί τώρα σχεδόν σε κάθε χώρα μέλος έχουμε διαφορετικούς κώδικες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σημαντικότατη ευθύνη για τους εθνικούς ρυθμιστές αλλά και για τον Ευρωπαϊκό, Οργανικό, για τον Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Οργανισμό, στο ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή. Επίσης το επίπεδο στήριξης των ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας πρέπει να είναι συνεκτικό. Είναι αδύνατο να υπάρξει εμπόριο, εμπορία δηλαδή ανανεώσιμων ε, πηγών, δηλαδή ε, ηλεκτρικού ρεύματος που έρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν έχουμε σε μια χώρα μια τεράστια υποστήριξη από το δημόσιο δηλαδή για τις ε, ε, πηγές αυτές και σε άλλη χώρα σχεδόν μηδενική. Είναι αδύνατο να γίνει, διότι τότε θα είναι σαν dumping. Άρα βήμα προς βήμα πρέπει να καταργήσουμε τα κίνητρα. Όχι μόνο για τα ορυκτά καύσιμα, για την πυρηνική ενέργεια, αλλά και στην περίπτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ίσως αυτό να ισχύσει μέχρι το 2020, αλλά το πιο υγιές για την αγορά ενέργειας θα, πρέπει να μην, θα, θα είναι να μην υπάρχουν κίνητρα για κανένα, για καμιά από τις πηγές ενέργειας. Και επίσης, να σταματήσουμε να ρυθμίζουμε τις τιμές. Δεν θα πρέπει να ρυθμίζουμε τις τιμές στις χώρες μέλη, τις τιμές ενέργειας. Γιατί και αυτό δεν είναι υγιές από την άποψη του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητάς μας και της θέσπισης του επίπεδου των τιμών ενέργειας. Θα πρέπει να θυμηθούμε πόσο ευάλωτη είναι η αγορά μας και ιδίως τμήμα των καταναλωτών που θα χρειάζονται πάντοτε βοήθεια, ίσως 12-15%. Οι υπόλοιποι όμως θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τιμές απολύτως ελεύθερες. Να είναι η αγορά φιλική στους χρήστες, όπως είπε και ο υπουργό Νεβερόβιτς. Τελευταίο επιχείρημα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε συντάξει πολλή νομοθεσία. Το τρίτο πακέτο ενέργειας, το πιο σημαντικό, του έτους 2009, του Μαρτίου, με τσεχική προεδρία τότε, όπου συμφωνήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαναλέω τον Μάρτιο του 2009, τότε ήταν η προθεσμία μέχρι το 2011 δηλαδή για την εφαρμογή προβλέπεται μια διετία και όσο γνωρίζετε 18 χωρίς μέλη δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα το πακέτο εκείνο. Και βεβαίως και πολύ άλλα σημαντικά νομοθετήματα. Τον κανονισμό για την ασφάλεια της προμήθειας αερίου. Πολύ, πολύ σημαντικός από την σκοπιά της ασφαλούς προμήθειας ε, αερίου. Επίσης για την πυρηνική ενέργεια. Επίσης, μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χωρών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας. Πολύ σημαντικό, πώς να ανταλλάσσουμε πληροφορίες δηλαδή για όλες τις διαπραγματεύσεις μας, έτσι ώστε να είμαστε ισχυρότεροι στις διαπραγματεύσεις με τους εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωση εταίρους και για την υποδομή κτλ. Πολύ σημαντική νομοθετική εργασία. Αγαπητέ φίλοι, αγαπητοί φίλοι, προέρχεστε από, χώρες, από διαφορετικέ χώρε μέλη. Είναι σημαντικό οι χώρε μα, οι κυβερνήσει μα, τα εθνικά μα κοινοβούλια θέλουν να εφαρμόσουν την νομοθεσία μα. Και πρέπει, γιατί αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία τη ενιαία μα αγορά. Η νομοθεσία υπάρχει, όλα έχουν κατατεθεί επιτάπητο και όμω δεν εφαρμόζονται ακόμη. Πρότεινα μαζί με τον Ζακ Ντελόρ, πρώην πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα είδος ευρωπαϊκής κοινότητας της ενέργειας. Προτριετίας ξεκινήσαμε μια πολιτική ιδέα. Πώς να συντάξουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική, όπως για παράδειγμα την κοινή αγροτική πολιτική, παρόμοια. Τρία χρόνια μετά, σχεδόν φτάσαμε να υλοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη ιδέα με την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα αυτό που χρειαζόμαστε κυρίως είναι η ρύθμιση και η εφαρμογή στις χώρες μέλη. Χρειαζόμαστε κάποια έξτρα προσπάθεια για διαμεθοριακές διασυνδέσεις καθώς και την εξέβρεση των απαραίτητων λύσεων για την ελεύθερη εμπορία της ενέργειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε, εφόσον επιτευχθούν αυτά, μπορούμε να αναμένουμε σταθερότητα τιμών, φθηνές ανταγωνιστικές τιμές και ταυτόχρονα προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Μπουζέκ για την παρέμβασή του που διαβιβάζει και το πάθος ε, με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Βιομηχανίας αλλά και δύο παρακολουθούν το θέμα αυτό. Τώρα, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Ο Επίτροπος Ετινκέρ έπρεπε να κυρώσει τη συμμετοχή του λόγω μιας αποστολής ε, της τελευταίας στιγμής, αλλά θα καλωσορίσω το Φίλιπ Λό, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένας διευθυντής ο οποίος πάντοτε ήταν παρόν στις εργασίες της Επιτροπής μας και πάντοτε έδινε και μεγάλη προσοχή στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, Φίλιπ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη, των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που ακούω από τον Επιτρόπο Έτιγκερ σήμερα το πρωί εδώ ουσιαστικά δεν μπορούσε να έρθει γιατί συμμετέχει στην υπογραφή του τμήματος του Νοτιού Διαδρόμου που είναι ένα μεγάλο ε, βήμα για την ε, εναλλαγή ενεργειακού εφοδιασμού να απομακρυνθούμε από τους παραδοσιακούς πραγματευτές μας. Ευχαριστώ την Λιθουανική Προεδρία και τον Πρόεδρο Σεμαϊτάκης ε, και την Πρόεδρο που οργανώσαν ε, αυτή τη συνάντηση. Ο διάλογος με τα Εθνικά Κοινοβούλια ποτέ δεν ήταν τόσο ουσιαστικό γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μεγάλη σύγκληση μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών στον τομέα της ανέργειας αν θέλουμε να πετύχουμε τους συνολικούς μας στόχους. Και θα έλεγα, Πρόεδρε, ότι αυτή η συζήτηση λαμβάνει χώρα σε μια πολύ κατάλληλη στιγμή. Ζητήθηκε από την Κομισιόν να παρουσιάσει προτάσεις τον Ιανουάριο για να προετοιμάσει δύο ευρωπαϊκά συμβούλια, ένα το Φεβρουαρίο για την ανταγωνιστικότητα και το δεύτερο για τις ενεργειακές τιμές και την αγορά ενέργειας και το μελλοντικό πλαίσιο μετά το 2020 και στο πλαίσιο της ε, κοινή μας συνεργασίας, ε, δηλαδή μεταξύ Συμβουλίου Κομισιών ε, και Κοινοβουλίου για το πλαίσιο μετά το 2020 είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τους στόχους που θέσαμε το 2008. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταγίδα γύρω από τις ενεργειακές πολιτικές και είδαμε και τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης η οποία ουσιαστικά έχει πλήξει τις επενδύσεις. Είχαμε τη Φουκοσίμα η οποία περιόρισε τις επιλογές που είχαμε στη θέση μας και έχουμε την επανάσταση του σχεσταθλητικού αερίου στις Ηνωμένε Πολιτείε και έχει αυξήσει το χάσμα μεταξύ Ευρώπης και ΙΠΑ και έχουμε αυξανόμενη ανησυχία σε όλες τις χώρες σε σχέση με την δυνατότητα να έχουμε φτηνή ενέργεια και τον αντίκτυπο των μισθών ε, που δεν αυξάνονται, ενώ έχουν αυξηθεί οι τιμές της ενέργειας, ε, κυρίως λόγω της ασιατικής αίτηση, για ορεικτά καύσιμα, αλλά και από άλλου παράγοντες. Αν ε, δούμε τώρα τους παραδοσιακούς στόχους του να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή και ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά της ενέργειας στην Ευρώπη, κυρίως την ηλεκτρική ενέργεια και τον αέριο, μπορεί να πει κανείς στο πλαίσιο αυτό ότι να ολοκληρωθεί αυτή η αγορά ενέργειας είναι μία επιλογή που δεν την ε, μετανιώνουμε ε, και ε, αυτό καλύπτει τα πάντα. Και αν θυμηθείτε το χάρτη πορείας που είχε εκπονηθεί για το 2050, που δεν ήταν στρατηγική, αλλά βασιζόταν επί της χάραξης οικονομικών μοντέλων, όπως είχε εξηγήσει η Κομισιόν, βλέπουμε ότι είναι πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε όπως και να έχει σε κάθε περίπτωση. Και ένα από αυτά είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα, περισσότερες ανανεώσιμες, έξυπνες υποδομές και ενεργειακή αποδοτικότητα αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και έχουμε καθήκον να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ε, για να ε, κάνουμε την ε, μετάβαση με το μικρότερο δυνατό κόστος, όπως είπε και ο κύριο και η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μπορεί να συνεισφέρει τα μάλα για την ανάκαμψη της οικονομίας γενικά. Και δεν είναι μόνο η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο που συμφωνούν επ' αυτού οι διαβουλεύσεις ε, κατόπιν ε, της πράσινης βίβλου της Κομισιόν ε, για το πλαίσιο 2030 για τις κλιματικές αλλαγές και τις κλιματικές πολιτικές δείχνει ότι υπάρχουν πολλά ωφέλη από την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και ισχυρή υποστηρίξη για περαιτέρω ολοκλήρωση της αγοράς παρά να επιτρέψουμε τον κατακαιρματισμό της αγοράς και η στρατηγική που υλοποιήθηκε από την Bush Consultancy μας ε, έδειξε ότι το κόστος της μη ολοκλήρωσης εσωτερικής αγοράς μπορεί να φτάσει ε, από τα 40 μέχρι τα 70 δισεκατομμύρια ετησίως, δηλαδή να μην έχουμε το όφελος του περαιτέρω ανταγωνισμού και της συγκράτησης των τιμών να μην μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τον εφοδιασμό με έναν αποτελεσματικό ως προς τον κόστος τρόπο για κάθε κυβέρνηση και για κάθε εταιρεία. Όποιοι στόχοι έχουν τεθεί για την περίοδο μετά το 2020 για το κλίμα θα πρέπει να επιτευθούν με ένα αποτελεσματικό πρωτοκόστος τρόπο και η εσωτερική αγορά αποτελεί προπόθεση γι' αυτό. Εμείς στην Κομισιόν βάζουμε τη δυνατά μας για να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα, λέγοντας στις κυβερνήσεις ότι έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν την νομοθεσία για την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά στην ενέργεια, επαναλαμβάνοντας τα οικονομικά επιχείρηματα υπέρ του να λειτουργεί η αγορά σε πανευρωπαϊκή βάση και η πανευρωπαϊκή διάσταση της ενεργειακής αγοράς θα πρέπει να μας ξεγελάσει στο να πιστέψουμε ότι αυτό ξεπηδά από το εθνικό επίπεδο και φτάνει αμέσως στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πιο σημαντικό για την εμπορία και την επένδυση στην ενέργεια είναι να βρούμε τις ευκαιρίες να το πράξουμε με τους άμεσους γείτονες γιατί ε, οι φυσικές συνδέσεις και ο συνδυασμός στόχων μαζί είναι κάτι ζωτικό και λίγοι που έχουμε ήδη αναπτύξει στην ε, αγορά αερίου θα πρέπει να επεκταθεί για να καλύψει και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, βασιστήκαμε στην νομοθεσία που έχουμε Ακούσαμε και τον κύριο Μπουζέκα και ανέφερε και άλλε πρωτοβουλίε αυτή τη Επιτροπή ε, και βασιστήκαμε σε αυτή την όθηση για να ολοκληρώσουμε και του κωδικού δικτύων. Χρειαζόμαστε όμω δημόσια στήριξη και για τι ανανεώσιμε πηγέ αλλά και για τι αγορέ χωρητικότητα και πρέπει να δούμε πώ οι τιμέ και το κόστο επηρεάζουν την ανταγωνιστική μα θέση. Επίσης να τονίσω ότι κάτι είναι ξεκάθαρο στο μελιώδης αρχή οι αγορές αν δεν είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο είναι τουλάχιστον ε, το λιγότερο ε, χειρότερο και αν χάσουν όσοι χαράσουν την πολιτική την πίστη τους σε αυτή την αρχή μπορεί να λαμβάνουν μέτρα που είναι αντιπαραγωγικά μακροπρόθεσμα και δεν ε, επιτρέπουν στην αγορά ε, να καταλήξει σε ωφέλη αποδοτικότητας. Θα παρουσιάσω κάποια παραδείγματα. Τα κράτη-μέλη καταρχήν πρέπει να δουν εκ νέου πώς παρεμβαίνουν στις αγορές. Η παρέμβαση και η στρέβλωση της αγοράς γίνεται σε διάφορα επίπεδα της ε, αλυσίδας αξίας με την προστασία των καταναλωτών με ρυθμισμένες τιμές χωρίς να Σημαίνει αυτό ότι δεν χρειάζεται κάποιο μεταβατικό στάδιο ε, στο μέγεθος των εκτόσεων για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τον αντίκτυπο αυτών των εκτόσεων για τους υπόλοιπους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και ε, κάποια συστήματα πολύ γενναιόδωρα ε, για ε, κάποιες νέες τεχνολογίες καθώς και οι επιδοτήσεις που δίνονται από το κράτος μόνο σε εθνικούς προμηθευτές. Τα μέτρα αυτά έχουν πολύπλοκα αποτελέσματα, συνήθως αρνητικά, αλλά το πιο σαφές από όλα είναι ότι έχουν πολύ σημαντικά διασυνοριακά αποτελέσματα εκεί όπου η ικανότητα διασύνδεσης είναι ήδη πολύ ψηλή. Θα πρέπει να δώσουμε χώρο να ανθίσει η εσωτερική αγορά. Ε, δεν θα πρέπει να την περιορίσουμε, πρέπει να επιλέξουμε όχι αποκλίνουσες εθνικές πολιτικές, αλλά συγκλίνουσες. Οι δύο υπουργό και ο πρόεδρο Μπουζίκα αναφέρθηκαν σε αυτό και θα το πω και εγώ. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε αποτυχία να εφαρμόσουμε πράγματα που έχουν συμφωνηθεί ευρέως ε, σε νομοθετικό επίπεδο στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Όταν κάτι έχει συμφωνηθεί θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι απαράδεκτο να ζημιώνουμε την εσωτερική αγορά αν δεν ε, μεταφέρεται στην εθνική νομοθεσία το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η Κομισιόν δεν θα διστάσει το να ξεκινήσει διαδικασία κατά ήταν να ε, καταπολεμήσει τις εθνικές επιδοτήσεις. Ε, το πακέτο που εθετήθηκε το 2009 υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο ιστορικό δίκαιο μέχρι το Μάρτιο του 2011. Ακόμη 12 ε, υποθέσεις κρεμούν 2,5 χρόνια μετά για μη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και στις δύο περιπτώσεις έχουμε οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επίσης αξιολογούμε τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία, καθώς πολλές κοινοποιήσεις έφτασαν πρόσφατα. Τώρα, δείτε τις τεράστιες ανάγκες σε επενδυτικό επίπεδο. Για να λειτουργεί η ενεργειακή αγορά, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ικανότητα παραγωγής και μεταφοράς ε, της ενέργειας ε, εκεί όπου δεν ε, λαμβάνουν χώρα οι επενδύσεις ή δεν λαμβάνουν χώρα με αποτελεσματικό τρόπο επειδή δεν έχουμε σαφές νομοθετικό πλαίσιο υπάρχουν προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει το επενδυτικό περιβάλλον με τη σταθερότητα που χρειάζεται. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις αρμοδιότητες της για να οθεί τα κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση της πληρούς εφαρμογής. Ένα σημαντικό στοιχείο της σημερινής συζήτησης, ωστόσο, θα συνεισφέρει στον να επικεντρωθεί η συζήτηση στην ανάγκη για ευρωπαϊκές λύσεις σε σχέση με τις τιμές. Εμείς προετοιμάζουμε μία πλήρη έκθεση, όπως είπα και νωρίτερα, για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, το Φεβρουάριο. Την περασμένη εβδομάδα, ο αρμόδιος οργανισμός για το συντονισμό των εθνικών συντονιστών, των εθνικών συντονιστικών αρχών ΕΣΑ, παρουσίασε μια έκθεση παρακολούθησης και τα συμπεράσματα είναι σαφή ότι οι τιμές στον τελικό καταναλωτή έχουν αυξηθεί και πάλι στην Ευρώπη το 2012, 45% για την ηλεκτρική ενέργεια και 10% για το αέριο. Χρειαζόμαστε πλήρη διαφάνεια για τους ε, λόγους ε, των εξελίξεων των τιμών. Χρειάζεται να αναλύσουμε τη διαδικασία σε διάφορες ε, συνιστώσεις ό,τι αφορά του φόρους, την ενέργεια, τους δεσμούς, Η Κομισιόν κάνει μια έρευνα τώρα. Η φορολογία και οι φόροι του δικτύου τώρα αποτελούν πάνω από το 50% ε, του λογαριασμού και είναι δυσανάλογη σχέση αυτή σε πολλά κράτη-μέλη. Τώρα, όσο πιο, πιο μικρή είναι αυτή η συνιστόσα, τόσο μικρότερη δυνατότητα για ανταγωνισμό έχετε εσείς ένα σημαντικό ρόλο στο να ελέγχετε την κατεύθυνση που ακολουθεί η πολιτική σε εθνικό επίπεδο και να επηρεάσετε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές και εθνικές πραγματικότητες. Ο Επίτροπος μου έχει πει πολλές ε, φορές ε, ότι άλλα λένε και άλλα κάνουν οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, με δύο λόγια, τα κράτη-μέλη είναι μεν θεωρητικά υποστηρίζουν τι αγορέ, αλλά μερικέ φορέ εμφανίζεται στην πράξη μια διαφορετική εικόνα. Αν πράγματι θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτε και τι επιχειρήσει από τι υψηλέ τιμέ στην ενέργεια, ο καλύτερο τρόπο, είναι να το κάνουμε όχι θέτοντα τις τιμές κάτω από την πραγματική αξία, αλλά διασφαλίζοντα ότι ε, μια εύρωστη λειτουργική αγορά μπορεί να παράσχει δικέ τιμέ. Η επενδυτές θέλουν υψηλότερε τιμές, οι καταναλωτέ χαμηλότερε τιμές και πρέπει να αφήσουμε την αγορά να κρίνει την αξία του τι απαιτείται και να δώσει κίνητρα ε, για τον εφοδιασμό που είναι απαραίτητο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Χλιλιπλό για την ε, παρουσίασή του. Τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση. Έχουμε πάρα πολλούς που έχουν ζητήσει το λόγο. Επομένως ε, πρέπει να σεβαστούμε αυστηρά το χρόνο ομιλίας. Έχουμε θέσει τους εξής κανόνες. Θα δίνουμε το λόγο σε δύο μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και κατόπιν σε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δύο, ένας, δύο, δηλαδή έτσι θα είναι η εναλλαγή. Και θα έχετε χρόνο ομιλίας δύο λεπτά για κάθε παρέμβαση. Ήδη 20 άτομα έχουν ζητήσει το λόγο, επομένως ας προσπαθήσουμε να σεβαστούμε το χρόνο. Όποιος ε, θέλει να πάρει το λόγο πρέπει να συμπληρώσει ένα έγγραφο που λέει Request for Speaking Time, έχει διανεμηθεί. Αν θέλετε μπορείτε να το συμπληρώσετε και να μας το παραδώσετε. Να ξεκινήσουμε καταρχήν ε, με τη συνάδελφο Μπριτε από τη Λιθουανία που είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Εθνικού της Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές. Ως ε, μέλος του Λιθονικού Κοινοβουλίου, με τα χαράς άκουσα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας στον τομέα της ενέργειας. Η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ε, στην ενέργεια είναι μία από τις κύριες προτεραιότητές μας και θα πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος για την επόμενη δεκαετία. Θεωρώ ότι μετά τα επόμενα δέκα χρόνια δεν θα πρέπει να παραμένουν άλλες ενεργειακές νησίδες στην Ευρώπη. Παρόλες τις προσπάθειες απελευθέρωσης ε, της αγοράς και παρά την υλοποίηση ε, του τρίτου πακέτου για την ενέργεια, την τελευταία δεκαετία οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί. οι καταναλωτές δεν συμμετέχουν πολύ, δεν είναι δραστήριοι στην αλλαγή παρόχου και οι πάροχοι δεν ενεργούν με διαφάνεια όταν αυξάνονται τις τιμές. Κατά τη διαπραγμάτευση των τιμών με τρίτες χώρες θα πρέπει να μιλάμε με μία φωνή. Ωστόσο, δεν πρέπει να πρόκειται μόνο για μια γενική δήλωση. Θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένους στόχους για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θέλουμε λοιπόν μεγαλύτερη συνέπεια σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική για το ε, συστολιθικό αέριο και πιο ενοποιημένη ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να διασφαλίσουμε και ανταγωνιστικές τιμές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Αγιατόγια, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ε, του Κωσοφοπεδίου. Παρακαλώ. Κυρία Σαρτόρη, εγώ θέλω να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος της Βουλής που καλέσατε την ε, Επιτροπή μας για να συμμετάσχουμε στη συζήτηση εδώ σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στις προκλήσεις και στα επιτεύγματα στο Κωσυφοπέδιο Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ακούμε για ενιαία ε, αγορά ενέργειας και για επενδύσεις και στις χώρες των Δυτικών ε, Βαλκανίων ε, ως μέλη της μελλοντική ενεργειακής αγοράς το Κωσυφοπέδιο αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα και προκλήσεις σε πολλούς τομείς και ένας από αυτούς ήταν και η ενέργεια καθώς ε, ήταν η παραγωγή ενέργειας, η διασύνδεση, τα συστήματα διαμετακόμισης ε, κτλ. Τώρα, έχουμε πετύχει την ιδιωτικοποίηση του συστήματος διανομής, αλλά μπορώ να σας πω ότι και η διαδικασία αυτή δεν ήταν και τόσο εύκολη. Πρόσφατα συνάψαμε μια συμφωνία με τη Σερβία για την ενέργεια και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ενεργειακή αγορά. Εγώ μπορώ να πω σε σχέση με το κοινοτικό κεκτημένο ότι κάθε νομοθεσία που έρχεται στο Κοινοβούλιο ελέγχεται αν συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο και στο ε, κανονιστικό μας ε, γραφείο νομίζω ότι θα πρέπει να αναπτύξει το γραφείο μας με καλύτερη συνεργασία μαζί σας για να αποφύγουμε διάφορα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν σύν το χρόνο προκειμένου το κοσυφοπαίδιο να προετοιμαστεί κατάλληλα για να αποτελεί ένα μέρος της μελλοντικής αγοράς ενέργειας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για το χαιρετισμό στα Ιταλικά. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Πιλάρ Δελκαστίγιο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη του πάνελ και ιδίως ε, τον εκπρόσωπο της Λιθουανικής Προεδρίας. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση που κυρίως απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή, στον κύριο Λόου. Επί της αρχής φαίνεται ότι η Κομισιόν πρόκειται να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό σε σχέση με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής και την κλιματική αλλαγή για τα τέλη του Ιανουαρίου έτσι μας έχουν ανημερώσει τουλάχιστον στην Επιτροπή μας. Πρόκειται για μια λευκή βίβλο ή για κάτι παρόμοιο. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, καθώς έχουμε αυτή τη συζήτηση τώρα, Πώς το σκέφτεστε, πόσοι θα είναι αυτοί οι στόχοι για την κλιματική αλλαγή, ένας, δύο, τρεις, μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία ήδη από τώρα, γιατί όλα αυτά σίγουρα θα έχουν και αντίκτυπο για τις διάφορες δυνατότητες πηγών ενέργειας. Ευχαριστώ, Πιλάρ. Ο κύριος Σταμενίτης τώρα, μέλος της Επιτροπής Εμπορίου. από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Κυρία Σαρτίνη, αγαπητοί εκπρόσωποι των Κοινοβουλίων, των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική αντιμετωπίζει σήμερα ένα σύνολο προκλήσεων. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ασφαλή ενεργειακά αποθέματα που θα δίνουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις να έχουν φτηνή ενέργεια. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα για την σταδιακή μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και μια μετάβαση σε ενέργεια φιλικότερη προς το περιβάλλον. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η απεξάρτηση από συμβατικές μορφέ ενέργεια, όπω ο άνθρακα, και για να πετύχουμε το στόχο η Ελληνική Προεδρία θέτει τρει ημερομηνίε ορόσημο. Συγκεκριμένα, η προθεσμία του 2014 για ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η προθεσμία του 2015, οπότε κανένα μέλος κράτος δεν θα πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από τα δίκτυα της Ευρώπης και η συμφωνία του 2015 για τη διεθνή κλιματική αλλαγή. Η εμπειρία της οικονομικής κρίσης έμαθε σε εμά τους Έλληνες ότι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ευημερίας των καταναλωτών, αλλά παράλληλα και της ε, προστασίας του περιβάλλοντος είναι η κατανάλωση ακριβής με υψηλό κόστος ενέργειας. Έχοντας την εμπειρία των τελευταίων χρόνων και γνωρίζοντας επιπτώσεις αυτού του φαινομένου, η προτεραιότητα που θέτει η Ελληνική Προεδρία στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής είναι εξή. Πρώτον, η επίτευξη των στόχων του 2020 για την ενέργεια και το κλίμα με την εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί γι' αυτό και δεύτερον η πρόοδο του πλαισίου πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το 2030 για να εξασφαλιστούν οι κατάλληλε επενδύσει που θα φέρουν βιώσιμη ανάπτυξη, για και ανταγωνιστικέ τιμέ ενέργεια με μεγαλύτερη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Διασφαλίζοντα ότι η έρευνα και η καινοτομία θα λειτουργήσουν για τη στήριξη των νέων στόχων. Κυρίως όμως θα ήθελα να προτάξω ότι από βασικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής είναι η διασφάλιση ότι το ενεργειακό σύστημα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα τη οικονομία Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας ανταγωνιστικές εγχώριες και διεθνές αγορές ενέργεια με τιμές που διεθνώς είναι ανταγωνιστικέ, προσιτέ στου καταναλ... τελικού καταναλωτέ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα νοικοκυριά και για τους παραγωγικούς κλάδους που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο ένα μέλος του Νορβηγικού Κοινοβουλίου. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Μία εύρυθμη λειτουργία της αγοράς συνδέεται με τις ε, διασυνδέσεις ε, στις φυσικές υποδομές. Ε, στις ε, χώρες Σκανδιναβίας έχουμε αυτή την εύρυθμη λειτουργία της ολοκληρωμένης αγοράς με διάφορα σημεία διασύνδεσης μεταξύ των χωρών μας. Αυτό μας επέτρεψε να έχουμε και κοινά πιστοποιητικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας. Και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό για την περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ Βάσει τη δική μα εμπειρία θεωρούμε ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προωθείται καλύτερα με τη διαμόρφωση αυτών των σημείων ε, διασύνδεση. Όμω, οι μηχανισμοί ικανότητα, όπω βλέπουμε ότι διαμορφώνονται σε διάφορα κράτη-μέλη, δημιουργεί στερβλώσει για την αγορά και μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την διαμόρφωση αυτών των interconnectors και για την ολοκλήρωση τη ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Η Νορβηγία ω χώρα παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια η ενέργειας μάλλον εν γέννη, μπορεί ε, να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια με την παροχή φυσικού ε, αερίου και υδροελεκτρικής ενέργειας. Όμως θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση ότι χρειάζονται ε, σημαντικές επενδύσεις εκ των προτέρων και έτσι απαιτείται οι σημαντικές ενδείξεις ενδιαφέροντος. Θα πρέπει λοιπόν όπως και να έχει να συμπεριλαμβάνονται οι interconnectors, αλλιώς τώρα που έχουμε δύο πολύ μεγάλα προγράμματα για τη Γερμανία και τη Βρετανία, για αυτά τα δύο προγράμματα λοιπόν θα υπάρξει ανασφάλεια, κάτι το οποίο θα αποβεί καταστροφικό για αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βιτόριο Πρόντι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο μεγάλη είναι η διάσταση του θέματος ε, της ευρωπαϊκής ενέργειας. Επομένως, ε, θα ήθελα να τονίσω ότι χρειάζεται να επενδύσουμε σε τεχνολογίες που να είναι ιδιαίτερα αποδοτικές στο θέμα της μεταφοράς και σε υψηλή τάση, συνεχή. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα δίκτυο το οποίο να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό και να μπορεί να, να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές αιωλικής ενέργειας και να μειώσουμε και την αναγκαιότητα αποθήκευσης της ενέργειας. Αυτή είναι μια ευρωπαϊκή υποδομή και εγώ νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να την υλοποιήσουμε με ευρωομόλογα και αυτό το συντομότερο δυνατόν. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω πως εμείς ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μεταξύ της ε, παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα από τη βιομάζα και με την αναγκαιότητα της ε, προστασίας του εδάφους λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η συνέργεια μπορεί να γίνει και να ωφελήσει και την ασφάλεια του εδάφους και τον ενεργειακό εφοδιασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Πρόντι. Τώρα το λόγο έχει Νεχάτ ε, Ζεμπέσκι, πρόεδρος ε, της Επιτροπής Τεχνολογίας και Φυσικών Πόρων από το Τουρκικό Κοινοβούλιο. olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας διαβάσω το χαιρετισμό του Τουρκικού Κοινοβουλίου. Θα προσπαθήσω να μιλήσω αργά στην Τουρκία, στον τομέα της ενέργειας. Όταν μιλάμε για το θέμα της κατανάλωσης, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ και θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα σημεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ε, κατανάλωση ενέργειας, ε, θα ήθελε οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν ενέργεια αξιόπιστη, φτηνή, σε λογικές τιμές και φυσικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, από όσο γνωρίζω, σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται σε ιδιαίτερο πλεονέκτημα η περιοχή της Κασπίας, η Ασία και η Μέση Ανατολή είναι οι περιοχές ε, που διαθέτουν ε, ενεργειακές πηγές, ενεργειακούς πόρους και επομένως προφανώς ε, η Τουρκία θα μπορούσε να αποτελέσει μια γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιοχών όπου βρίσκονται αυτοί οι φυσικοί πόροι. Και γι' αυτό το λόγο η Τουρκία σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την καταναλώση θα μπορούσε να λάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Τα τελευταία 11 χρόνια βλέπουμε ότι η κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 1,6% ενώ στην Τουρκία βλέπουμε ότι το νούμερο αυτό έφτασε στο 5% και τα επόμενα 10 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2022 η Τουρκία θα πρέπει να πολλαπλασιάσει ε, τα νούμερα αυτά, γιατί όπως ξέρετε σημειώνονται ρυθμοί ανάπτυξης στην Τουρκία. Η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μέλος Όμως έχουμε προβλήματα με τη Βόρεια Κύπρο. Η Βόρεια Κύπρος είναι απομονωμένη και είναι σημαντικό όταν μιλάμε για ολοκλήρωση η ολοκλήρωση να μπορεί να γίνει ολοκληρωμένα. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην εκπρόσωπο της Βουλής των Λόρδων που προέρχεται από την Επιτροπή, στην κυρία Σκότ, προέρχεται από την Επιτροπή Ελίας και Γεωργίας. Ευχαριστώ, καλημέρα. Το Μάιο φέτος ε, η Επιτροπή της οποίας προεδρεύω δημοσίευσε μια έκθεση για την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης ε, για την αποφυγή ακριβώς την απαλυφή αυτών των ε, εικονισίδων. Και χαίρομαι που ε, αυτό αναφέρθηκε και από τους ε, σημερινούς ομιλητές, ιδίως ό,τι αφορά τη σημασία της διασύνδεσης και της ολοκλήρωσης της εσωτερική αγορά. Όμω, η βασική πρόκληση την οποία εμεί εντοπίσαμε στην έκθεσή μα είναι η πρόκληση των επενδύσεων. Χρειαζόμαστε επενδύσει ενό τρει μέχρι το 2020 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρόσφατα έγινε ένα σεμινάριο στο Λονδίνο, στο City, για να απευθυνθούμε στου επενδυτέ για αυτό το ζήτημα. Το καλό είναι ότι υπάρχουν ε, πολλά τρει που είναι διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο, όμω αποτρέπονται οι ε, επενδυτέ από την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ενεργειακό τρίλημα είναι ένα, μια γνωστή έννοια πλέον. Όμως ε, το βασικό είναι η βεβαιότητα, η ασφάλεια αφορά φορά τις ε, τιμές ε, και την ε, προμήθεια της ενέργειας. Γιατί ακόμα και αν έχουμε κάποιου βραχυπρόθεσμου στόχου, αυτό θα πρέπει να αποκατασταθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Και αυτή η ασυμβατότητα είναι που αποτρέπει του επενδυτές. Για παράδειγμα, ο, ανανεώσιμος, ο στόχος για τι ανανεώσιμε μέχρι το 2020 ήταν πολύ επιτυχής για την προώθηση των επενδύσεων σε αυτό το τομέα. Όμως, πέραν το 2020 έχει πέσει η εμπιστοσύνη και σίγουρα... Ε, ε, θα πρέπει να πάμε πέρα από του στόχου μείωση των εκπομπών άνθρακα. Και τέχω, τέλος ε, δηλώνουμε ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ε, τοπική διανομή ε, της ενέργειας και στην παροχή κινήτρων για την αύξηση των καταναλωτών. Ευχαριστώ κυρία Γκέμπελς. Κύριος Γκέμπελς, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Όταν η Επιτροπή εκκίνησε αυτή τη διαδικασία της ολοκλήρωσης αγοράς, μας είχε υποσχεθεί ότι θα πέσουν οι τιμές. Είναι σαφές ότι αυτό δεν έγινε. Τώρα ο Φίλιπ Λό μας είπε ότι όταν θα ολοκληρωθεί η αγορά, τότε θα πέσουν οι τιμές. Δεν ισχύει αυτό. Και οι λόγοι είναι απλοί. Πρώτον, έχει μειωθεί ο ανταγωνισμός. Γιατί ε, κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις είναι σε περισσότερε εθνικέ αγορές. Δεύτερον, οι καταναλωτέ δεν έχουν διαπραγματευτική ισχύ. Είναι όμοιροι. Ακόμα και οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις δεν έχουν διαπραγματευτική ισχύ εναντί αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων. Σίγουρα εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθούμε να κρυφτούμε από την πυρηνική ενέργεια, από το συλλογιστολιθικό ε, αέριο, ακόμα και για τα βιοκαύσιμα, είχαμε συζητήσεις και το καθεξής. Όμως ο βασικός λόγος είναι ότι δεν, η αγορά ενέργειας δεν είναι σαν τις υπόλοιπες αγορές. Τα 9 δέκατα της ενέργειας στον κόσμο πωλείται μέσω οντοτήτων που ελέγχονται από το κράτος. Τα 9 δέκατα των ε, συμβάσεων είναι ε, συμβάσεις μεταξύ κρατών. Και αυτό που συμβαίνει στις ε, spot markets είναι ακριβώς μια κερδοσκοπία, τίποτα παραπάνω. Κάθε τάνκερ πωλείται δεκάδες φορές πριν εξαχθεί κάπου. Δεν υπάρχει λοιπόν πραγματική ελεύθερη αγορά, υπάρχει αγορά που κυριαρχείται από μια χούφτα ε, επιχειρήσεων και ό,τι και αν ιδιωτικοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση δεν θα έχουμε καλύτερη λύση για τους καταναλωτές μας. Και το πρόβλημα στην κοινωνία μας είναι ότι έχουμε όλο ένα και περισσότερους ενεργειακά φτωχούς, τους οποίους θα πρέπει να επιδοτήσουμε αν θέλουμε να επιβιώσουν. Δεν έχω παραπάνω χρόνο για να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Μάνιος Μπρούνερ, μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ και για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, καθώς και για την πρωτοβουλία της ε, Λιθουανικής Προεδρίας. Τρία, τρεις παρατηρήσεις. Πρώτο, συμφωνώ ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να ξεφύγουμε από τις επιδοτήσεις, τα είπατε και εσείς από το πάνελ, πρέπει να τις εγκαταλείψουμε διότι στόχος κάθε επιδότησης δεν μπορεί να είναι άλλος παρά να φέρει σε επίπεδο οριμότητας μια νέα τεχνολογία. Βέβαια έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν και το κάρβουνο και η ατομική ενέργεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαφορετικές ταχύτητες εγκατάλειψης των επιδοτήσεων για να δώσουμε και στις ανανεώσιμες ενέργειες στην Ευρώπη μια δυνατότητα να επιβιώσουν και να καταφέρουμε να αλλάξουμε και την πορεία της ενέργειας σε ορισμένες χώρες. Σε ό,τι αφορά την υποδομή, πράγματι χρειαζόμαστε επιγόντως τις απαραίτητες υποδομές και κυρίως τις γραμμές υψηλής τάσεως που είναι σημαντική και για την στροφή, την αλλαγή στην ενέργεια διότι το ρεύμα παράγεται από τις ε, ανεμογεννήτριες και όταν ακόμα δεν τις χρειάζεται, δεν το χρειάζεται ο καταναλωτής. Την έχετε για παράδειγμα. Εκεί πρέπει να περάσουν λοιπόν να περάσει το ρεύμα με γραμμές υψηλές τάσους, πρέπει να περάσει και από τις Άλπεις. Εκεί χρειάζεται λοιπόν πολύ ε, υψηλό επίπεδο δαπανών επενδύσεων. Σε ορισμένε χώρε γίνεται συζήτηση επί δεκαετίε για το αν χρειάζονται γραμμές τάσεω των 380 kV. Επίσης, τίθεται και το λεγόμενο unbundling. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Δηλαδή, πρέπει η παραγωγή να ξεχωριστεί από τη διαχείριση του δικτύου διανομής. Δεν υπάρχει θέμα εκεί. Νομίζω όμως ότι όλες ρίχνεται όλες τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη στο ίδιο καλάθι, από την μικρή τοπική επιχείρηση μέχρι την πολύ μεγάλη. Και αυτό καμιά φορά οδηγεί σε πολύ παράδοξα αποτελέσματα, με συνέπεια πολύ σημαντική γραφειοκρατία που τελικά αποβαίνει σε βάρος των επιχειρήσεων αυτών. Και εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθίσει να σκεφτεί κάπως διαφοροποιημένες ρυθμίσεις για το κάθε είδος επιχειρήσεως. Ευχαριστώ τώρα ο κύριος Παμπλός Μάτος Μασκαρενιό, ο οποίος προέρχεται από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με τους στόχους, δηλαδή να πετύχουμε την εσωτερική αγορά ενέργειας. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο για την ασφάλεια εφοδιασμού όλων των κρατών, για τη βελτίωση των τιμών και για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε και ο πρόεδρος Μπούζεκ, δηλαδή στην ε, βελτίωση της εκβιομηχάνησης της Ευρώπης και όλων των κρατών μελών. Γι' αυτό είναι απολύτως ε, απαραίτητο να βελτιωθούν οι τιμές και να έχουμε όσο δυνατόν χαμηλότερες τιμές ενέργειας και είναι απολύτως απαραίτητο, αναμφισβήτητο, να βελτιωθούν οι διασυνδέσεις. Εμείς αξιολογήσαμε θετικά την έγκριση του πρώτου καταλόγου των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, των PCI, στους οποίους αναφέρθηκε ο κ. Σνοβέροβη. Πιστεύουμε όμως ότι δεν θα επιτευχθεί όλος ο στόχος του 10% για την ηλεκτρική ενέργεια στην προθεσμία που έχει προβλεφθεί. Επομένως, θεωρούμε ότι πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια χρηματοδότησης από την κοινωτική πλευρά προς όλες τις χώρες που αυτή τη στιγμή είναι ενεργειακές νησίδες. Και σε σχέση τώρα με τις τιμές, ε, είναι σημαντικό και αναφεσβήτητο το θα μπορούσαν να κατέβουν οι τιμές στην ιστορική αγορά, όμως πρέπει να αναλύσουμε ποιες είναι οι καθοριστικές, τι ε, είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για τις τιμές σε κάθε κράτος μέλος και όχι μόνο πρέπει να είναι ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία εναντί τριών χωρών, αλλά αυτό είναι σημαντικό και για την βιομηχανία των ίδιων των κρατών μελών για να ανταγωνιστούν και μεταξύ τους. Και εμείς είδαμε ότι ε, έχουμε το κόστος το χρηματοοικονομικό σε μια βιομηχανία και δεν χρηματοδοτούνται όλες οι χώρες με το διαπιτόκιο και έχουμε και το εργασιακό κόστος αλλά και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και προκειμένου να μπορούμε να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητα εντός της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει αυτό το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας να είναι παρόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Ρωμάνα Τζόρνταν. Παρακαλώ. Eh, ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Πρόεδρο και τον Πρόεδρο της Λιθουανικής Προεδρίας και έχω την εξής ερώτηση. Πώς βλέπετε την περαιτέρω εξέλιξη της ενιαίας αγοράς. Το τέταρτο πακέτο απελευθέρωσης έχει τώρα εγκριθεί, διότι το τρίτο αποδείχθηκε ανεπαρκές. Και με κάθε νέο πακέτο μιλούμε βεβαίως και για νέα εκχώρηση εθνικών αρμοδιοτήτων από τα Εθνικά Κοινοβούλια δηλαδή στις Ευρωπαϊκές Αρχές. Αυτό που θα ήθελα εγώ να γνωρίζω και απευθύνω το ερώτημά μου στους ε, βουλευτές των Εθνικών Βουλών, αν αυτοί θεωρούν ότι χρειαζόμαστε ακόμα πιο εναρμονισμένους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις επιδοτήσεις των ανανεώσιμων. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο στην παραγωγή των ανανεώσιμων. Χρειάζεται να ικανοποιηθούν επίσης και κάποιες νέες απαιτήσει ό,τι αφορά την αποθήκευση της ενέργειας. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αντί να υπάρχουν 27 ε, ξεχωριστές εθνικές αγορές. Επίσης, σε ποιο επίπεδο θα ήθελα να ρωτήσω, πρέπει να αναπτύξουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές πηγές ενέργειας. Δηλαδή, έχουμε τώρα αποκλήσεις απόψεων μεταξύ, για παράδειγμα, Γερμανίας και Ενωμένου Βασιλείου σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια. Η γερμανική απόφαση, άλλωστε, σημαίνει και κάποια τεχνικά προβλήματα για την ε, κυκλοφορία της ενέργειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τώρα και το στόχο του 2030, όπως εξήγησε ο κύριος Λόου προηγουμένως. Θέλω να μάθω όμως εσείς, οι εθνικοί βουλευτές, τι είδους ενεργειακές πολιτικές θεωρείτε ότι πρέπει να αναπτύξουμε μέχρι το 2030, στην περίοδο δηλαδή πρώτα μέχρι το 2020 και μετά μέχρι το 2030. Ποια πράγματα από αυτά που έχουμε κάνει θεωρείτε ότι ήταν ορθά και ποια όχι. Θα ήθελα να μάθω επίσης και για τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς αγοράς, για παράδειγμα το σύστημα εμπορίας εκπομπών ε, των αερίων του θερμοκηπίου και για τους τρεις στόχους, δηλαδή μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, αύξηση του επίπεδου ανανεώσιμων και πιο αποδοτική χρήση ενέργειας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιβαν Στράνσλαφ έχει τώρα το λόγο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Mm, Ευχαριστώ. Οι στόχοι της Πολωνίας συμπίπτουν με τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταγωνιστικότητα, ασφαλεία του φαδιασμού και βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτοί οι τρεις κοινοί στόχοι. Όπως είπε ο κ. Μπούζεκ, το σημαντικό είναι η ανταγωνιστική αγορά που είναι και για μας κάτι σημαντικό. Και αυτό έχει να κάνει με τις διασυνδέσεις, ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των υποδομών. Αυτό περιλαμβάνει και την ανάπτυξη των υφείων δικτύων. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας στο να χρησιμοποιήσουμε την τοπική ικανότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα θέμα που άπτεται της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Η Πολωνία, όπως ε, και άλλα κράτη-μέλη, μπορεί ελεύθερα να επιλέξει το ενεργειακό της μείγμα. Εμείς θα συνεχίσουμε να, να χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνολογιών, ε, αλλά ο άνθρακας ε, θα παραμείνει σε μεγάλη χρήση τα επόμενα έτη. Επίσης θα χρησιμοποιούμε περισσότερο φυσικό αέριο, καθώς θα ανοίξει και ένα θερματικός σταθμός στο Σφινόιτσι και επίσης θα εφοδιαζόμαστε και από την Κροατία. Θα έχουμε λοιπόν και δύο εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού αερίου. Τώρα, αυτό το ενεργειακό μείγμα είναι ε, κάτι το οποίο αποφασίζεται από τους επενδυτές μας. Επομένως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε στο στόχαστρο και τους καταναλωτές. Ορισμένες από την ανασιώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα και εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 θα έχουν καταστεί ανταγωνιστικές. Κατανοούμε λοιπόν την ανάγκη να υπάρξουν επιδοτήσεις για αυτές τις πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διαφορετικά θα δούμε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Και το αποτέλεσμα θα είναι να μην έχουμε ανταγωνιστική αγορά. Επίσης, ε, θέλουμε να επικεντρωθούμε στις ε, πολιτικές σχετικά με την αλλαγή του κλίματος μετά το 2030. Στα πλαίσια των πολιτικών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αν δούμε και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, είναι κάτι πολύ σημαντικό και η καθαρή τεχνολογία είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Πολωνία. είναι μια πολύ σημαντική πηγή ενέργειας αυτή και για την Πολωνία και για άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ζητώ να σεβαστείτε το χρόνο για να μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο. Διαφορετικά, αν ε, όλοι μακρηγορήσουν τόσο πολύ, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όσους τον έχουν ζητήσει. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κρίστινα Κικικύρου, ο οποίος είναι μέλος της ε, Οικονομικής Επιτροπής για τη Βιομηχανία και τις ε, Επενδύσεις της Ρουμανίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρου ε, τη ε, Ρουμανική Γερουσία θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παρευρεθούμε εδώ σήμερα σε αυτή την ε, τόσο κρίσιμη σημασία συνεδρίαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι και η Ρουμανία θέλει να βρει λύσει για να διασφαλίσει την ενεργειακή τη ανεξαρτησία, θα ήθελα εδώ να πω ότι έχουμε δύο σημαντικές προκλήσεις για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια φοδιασμού στο φυσικό αέριο της Ρουμανίας. Α, συγγνώμη, λέει ο μιλητής. Και η δεύτερη πρόκληση για τη Ρουμανία είναι ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα υδροελεκτρική ενέργεια. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να θέσω τρία ερωτήματα προ τον ε, κύριο Γενικό Διευθυντή. Πρώτον, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ε, ρύθμισης των τιμών της ενέργειας. Θα υπάρξει καθεστώς στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τι πρόοδος έχει σημειωθεί για την κατάλληλη αξιολόγηση των κινδύνων εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού αερίου στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντρες Περέα, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την οργάνωση αυτής της συζήτησης. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε. Όμω εγώ θέλω να θέσω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο Κομισιόν. Μα είπε ότι οι κρατικέ ενισχύσει τρευλώνουν την αγορά και πράγματι το πιστεύω και εγώ. Γιατί έχουμε μέχρι και νέα υποθέσει που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Ε, μπορείτε να μα πείτε ποιε είναι αυτέ οι υποθέσει, να τι απεριθμίσετε. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της Κομισιόν για την ενιαία αγορά ενέργειας ε, και ποια θα είναι η βαρύτητα των ανανεώσιμων δηλαδή να μας ε, πείτε η Κομισιόν ε, ποιο είναι το βάρος που δίνει σε νέες πηγές ενέργειας ε, για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπρέα. Τώρα θα δώσω το λόγο στο κύριο Ράτα, ο οποίος είναι πρώην συνάδελφος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Σλοβακίας. Παρακαλώ. Έχω ξεχάσει λίγο πώς λειτουργεί. Ευχαριστώ λοιπόν που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Πρώτα εκφράζω τις ευχαριστίες μου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προχώρησαν τόσο πολύ για την ολοκλήρωση της ε, ενιαίας αγοράς ενέργειας και να βοηθήσουν να ξεπεραστεί αυτή η ενεργειακή απομόνωση τόσων χωρών. Θα θυμάστε τη 2008-2009 την κρίση ενέργειας όταν σταμάτησαν οι εισαγωγές από τη Ρωσία, δηλαδή διέκοψε η Ρωσία τις εξαγωγές προς ε, τις ανατολικές χώρες της Ευρώπης το ε, φυσικό αέριο. Πρέπει στο μέλλον να φροντίσουμε να αποφευθούν τέτοιες καταστάσεις. Βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα τα κοινά έργα. Η Σλοβακία συμμετέχει αφενός στην διασύνδεση με αγωγούς φυσικού αερίου με Ουγγαρία και Πολωνία, καθώς επίσης με την Ουγγαρία πάλι για την μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος. Βρίσκω λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ευρωπαϊκά όργανα συμμετέχουν για τη δημιουργία αυτών των διασυνδέσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο εναρμόνισης της έννοιας ε, αγοράς ενέργειας. Θέλω να αντιδράσω στο ερώτημα της κυρίας Τζόρνταν που ζήτησε από εμάς, τους εθνικούς βουλευτές δηλαδή, να απαντήσουμε τι πιστεύουμε για την εναρμόνιση των κανόνων για τις επιδοτήσεις και για τα ορυκτά καύσιμα αλλά και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενέργειας. Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να εναρμονίσουν τους κανόνες αυτούς, διότι οι εθνικοί ρυθμιστές συχνά δεν βρούν όπως θα έπρεπε. Πρέπει να μειώσουμε βεβαίως αφενός τις κανονιστικές ρυθμίσεις, αλλά από την άλλη μεριά να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών, ώστε να είναι διαφανείς οι τιμές της ενέργειας και έτσι οι επιχειρήσεις μας να μπορούν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ ο κύριος Λίνα Μπάλσης ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αποδοτικότητα της αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο στο, από το πόσο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσει αποφάσεις όταν αν θέλει να επενδύσει ε, στις, ε, στα παροχημένα ορυκτά κάψωμα, κάψιμα ή στα πολλά υποσχόμενα ανανεώσιμα μέσα παραγωγής ενέργειας. Οι επιδοτήσεις προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να διαψεύσουμε το μύθο ότι υπάρχουν και τόσο τεράστιες επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες. Εάν η ηλιακή ή αιωλική ενέργεια ε, λάβει στήριξη, μέσα σε μερικά χρόνια θα ε, παράγει την ε, πιο αποδοτική ενέργεια. Αυτό το είδαμε και από τη Δανία. Νομίζω ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο μοναδικός τομέας που θα μας διασφαλίσει την ενεργειακή ανεξαρτησία και την ασφάλεια εφοδιασμού. Ας αποφασίσει ο κόσμος, λοιπόν, οι πολίτες τι είδους ενέργεια θέλουν στο μέλλον. Είχαμε δημοψήφισμα στη Λιθουανία κατά της πυρηνικής ενέργειας και ελπίζω να μην ε, ε, οικοδομηθεί αυτό το νέο πυρηνικό εργοστάσιο. Θα πρέπει να επενδύσουμε στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας. Κάθε κτίριο ή επιχείρηση να έχει τις δικές της εγκαταστάσεις ηλιακή ενέργειας. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει την οδηγία για την αποκατάσταση της ενέργειας που ε, παράγεται από τα νοικοκυριά. Και για τα ευφύ δίκτυα θα πρέπει να τα στηρίξουμε γιατί τελείως θα υπάρχει διασύνδεση και δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αποδοτικά τις ανανεώσιμες μας. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε, να καταπολεμήσουμε τα λόμπι που είναι ιδιαίτερα δραστήρια σε ό,τι το σχιστολιθικό αέριο και τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό ο κλάδο βιομηχανία επιτέλου κατάλαβε ότι οι ανανεώσιμες πηγές Ενέργεια είναι πολύ φτηνέ και αποδοτικέ ε, πηγέ ενέργεια και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τι καταπολεμήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα το θα πάρει το λόγο ο κ. Τζον Λουκά Μπεραμάτι, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Δραστηριοτήτων, Εμπορίου και Τουρισμού από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί νομίζω ότι εδώ αναδύθηκε ένα από τα θέματα που ενδιαφέρει και πάρα πολύ τη χώρα μου. Η απέτηση για μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας για μας είναι απαραίτητη η αναγκαιότητα και εντός της κρίσης θα πρέπει να δώσουμε ανταγωνιστικότητα δυνατότητα ανταγωνιστικότητα στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Ε, τώρα θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια για τα δύο θέματα που συζητούμε. Το θέμα των υποδομών ε, και τη διασύνδεση αλλά και των κανόνων είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, για την υποδομή και την δυνατότητα Σύνδεση είναι ένα θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη και την ε, ικανότητα περιφερειακής παραγωγής που υπάρχουν σε διάφορες χώρες στην Επιρώ μας. Υπάρχουν χώρες που έχουν υψηλές δυνατότητες ανανεώσιμες ε, πηγε, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά χώρες όπως η δική μου χώρα που έχουν δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε, όπως θα πρέπει να σκεφτούμε και το στρατηγικό χαρακτήρα του εφοδιασμού. Εδώ ε, μιλήσαμε υπέρ του ανοίγματο του νοτιού διαδρόμου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε και τα αποθέματα που σιγά σιγά ανακαλύπτονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Χρειάζεται να εφαρμοστεί ταχύτατα το τρίτο πακέτο για την ενέργεια με ελεύθερη πρόσβαση στις εθνικές αγοράς. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσουμε ζωή στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας που να είναι ανταγωνιστική και να ε, θέσει ίδιους κανόνες για όλους. Και κάτι τελευταίο, μια τελευταία σκέψη αυτή τη στιγμή, ενώ καθορίζουμε τους ε, στόχους που θα θέσει η Ευρώπη για το 2030, πρέπει να ξέρουμε ότι οι στόχοι αυτοί δεν θα επιτευχθούν χωρίς ανισορροπίες αν δεν ε, θα έχουμε υλοποιήσει για εκείνη την περίοδο μια ισχυρή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Ευχαριστώ. Ο κύριος τώρα Ίγκορ Ραντάνοβιτς πρόεδρος της ε, Οικονομικής Επιτροπής της κρατίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερος για τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει και βεβαίως και για τις επιτυχίες που σημειώσατε με την υιοθέτηση του τρίτου ενεργειακού πακέτου καθώς και για όλα τα επιτεύγματα της Λιθουανικής Προεδρίας. Παρόλο που έχουμε μπροστά μας πολλά ανοιχτά ερωτήματα για τα οποία μίλησαν ήδη και συνάδελφοι από τη Σλοβενία και άλλες χώρες, παρόλα αυτά συμφωνώ με την γνώμη των μελών του πάνελ ότι αυτό το μέγα καθήκον που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή η ανάπτυξη των υποδομών για αυτή την ενεργειακή επανάσταση σημαίνει για μας σημαντική πρόκληση. Βέβαια, αυτό όπως είπε και ο πρόεδρος Μπούσεκ το χρειαζόμαστε για την οικονομική μας και βιομηχανική μας ανανέωση, που δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτή την ενεργειακή μεταρρύθμιση. Είναι βέβαια απαραίτητα σημαντικό και τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέψουμε, αλλά βεβαίως και να εξασφαλίσουμε την διανομή σε ολόκληρη την επικράτεια της ενιαίας αγοράς. Και χαίρομαι που δεν λαμβάνετε υπόψη σας μόνο τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις χώρες με τις οποίες παραδοσιακά έχουμε σχέση με τις χώρες δηλαδή της Ανατολικής Γειτονίας καθώς και των Δυτικών Βαλκανίων. Γι' αυτό και χαίρομαι που μπορώ να θυμίσω σήμερα ότι ιδιαίτερα στο Μπακού γίνεται σήμερα μια μεγάλη συνάντηση που ε, συζητεί την εναλλακτική επιλογή του Νότιου Αγού. Στην συνάντηση αυτή στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν συμμετέχουν και εκπρόσωποι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίοι προτίθεται να συζητήσουν και ενδεχομένως να υπογράψουν συμφωνία αμοιβαίας κατανόησης για την διανομή της ενέργειας και στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταβίντε Κρίκπε αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Παραγωγικών Δραστηριοτήτων από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας και για τη συζήτηση αυτή. Γιατί όταν μιλάμε αναλυτικά για θέματα, πραγματικά Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω από την υπερβολική παραγωγική ικανότητα που αφορά τη δική μου χώρα, αλλά και κυρίως ε, πολλές άλλες χώρες. Πώς θα διαχειριστούμε την ε, υπερβολική ικανότητα παραγωγής στα κράτη-μέλη. Σήμερα στην τελεία έχουμε δύο φορές την ικανότητα παραγωγής από αυτή την που είναι απαραίτητο. Αυτό νομίζω ότι θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ποιο θα είναι το κριτήριο της επιλογής, απλώς θα είναι οικονομικού χαρακτήρα ή θα αξιολογήσουμε ποιες είναι οι εκπομπές δεξιδίου του ένθρικα των μεμονωμένων συστημάτων παραγωγής ή του περιβαλλοντικού αντικτύπου τους. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο για να το συζητήσουμε και για να δώσουμε έναν ορίζοντα προοπτικών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της επίτευξης ε, των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο θέμα αφορά την κεντρική παραγωγή και τη διανομή της. Η ευρωπαϊκή πολιτική οδεύει προς τα εφη δίκτυα ε, και προς ένα σύστημα μικρών εγκαταστάσεων που θα είναι σκορπισμένα στην επικράτεια. Δεν κατανοώ πώς θα γίνει αυτό ε, όταν έχουμε σήμερα ένα σύστημα συγκεντρωτικό, δηλαδή έχουμε μεγάλες εγκαταστάσεις αυτά τα ευφυή e e δίκτυα ή αυτές οι e ευφυείς πόλεις θα μείνουν κατά κάποιο τρόπο θεωρητικές ιδέες. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μία παραγωγή και που θα διανέμεται και τοπική κατανάλωση της ενέργειας. Όχι να έχουμε ένα σύστημα μαζικής πώλησης ενέργειας το οποίο μας κάνει να πιστοχωρούμε πίσω στον χρόνο. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Τζενούπα Πασαϊσίτη από την Επιτροπή Ανάπτυξης Εμπορίου και Βιομηχανίας ε, από το Κωσυφοπέδιο. Παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό για μας σήμερα να γίνει, να σας πούμε μερικές με λεπτομέρειες και πληροφορίες ακόμα για εμάς, καθώς δεν είμαστε ακόμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοσφοπέδιο εξακολουθεί να δίνει μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη ε, ελεύθερης αγοράς ε, στον τομέα της ενέργειας. Έχουμε υιοθετήσει μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων για τη δημιουργία νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ε, ενεργειακή αγορά, την ανάπτυξη προγραμμάτων και τη στήριξη περιφερειακών προγραμμάτων και πρωτοβουλειών. Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό κλάδο και την αντίστοιχη νομοθεσία, να σας ενημερώσω ότι ήδη έχουμε υιοθετήσει έξι νομοθετήματα για την ενέργεια, Με την ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, για τη ρυθμιστική αρχή, φυσικό αέριο, ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή πολιτική στις επιχειρήσεις. Επιπλέον υιοθετήσαμε ρυθμίσεις, νομοθετήματα, διοικητικές διαδικασίες, μεθοδολογίες, Όλα αυτά από την κυβέρνηση και τα συναφή Υπουργεία. Για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Νομοθεσία να σας ενημερώσω ότι έχουμε εναρμονιστεί με το δεύτερο πακέτο για την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνει εύρωστη βάση για την αναδιάρθρωση του ενεργειακού κλάδου, κυρίως ό,τι φορά τον άνοιγμα της αγοράς και της αύξησης του ανταγωνισμού. Με την νομοθεσία μας έχουμε επιλύσει και άλλα σημαντικά ζητήματα για, τον, για το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού, της προώθησης της ενέργειας, της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Έχουμε υιοθετήσει και ενεργειακή στρατηγική και όλα όσα γίνεται αυτή τη στιγμή στο Κοσμοπέδιο βασίζονται ακριβώς σε αυτήν την ενεργειακή στρατηγική. Ευχαριστώ. Και η τελευταία παρέμβαση από τον κύριο Άντικε Κόνεν, που είναι μέλος της Επιτροπής Εμπορίου από τη Φιλανδία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στη διανομή Τη ηλεκτρική ενέργεια και τη ιδιοκτησία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει τάση δημιουργίας μονοπωλίων και ο πελάτης, ο καταναλωτή ουσιαστικά πρέπει να πληρώσει χωρίς να πει κουβέντα. Αυτό παρατηρούμε σήμερα. Το ερώτημά μου λοιπόν προς ομιλητές είναι θεωρείται σημαντικό το θέμα της ιδιοκτησίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα έπρεπε να είναι δημόσια, ιδιωτικά Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Υπάρχει διαφορά αν υπάρχει εθνική ιδιοκτησία του δικτύου ή ε, το δίκτυο ανήκει σε άλλη χώρα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και χώρα εκτός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα τις δικές σας απόψεις επί του θέματος. Αυτό ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε εδώ με τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρόνο. Και έτσι μπορούμε τώρα να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές για κάποιες απαντήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τον Υπουργό Νεβέροβιτς. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως ε, για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ακούσουμε τις απόψεις των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιβεβαιώνουν ακριβώς την κατεύθυνση στην οποία κινούμεθα. Ότι δηλαδή η ενοποίηση των εθνικών συστημάτων ενέργειας σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα είναι η κατάλληλη κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, για τα όσα είπατε ε, Αυτό είναι ο τρόπο που θέλουμε κι εμεί να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό και την ε, αποδοτικότητα στι ε, τιμέ τη ενέργεια και στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο για τα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει. Και σίγουρα θα τα εξετάσουμε όλα αυτά που είπατε, καθώ προχωράμε στο πιο σημαντικό στάδιο που είναι η υλοποίηση. Ακούσαμε από εσά ότι είναι ακριβώ πολύ σημαντική αυτή η υλοποίηση των όσων έχουμε επιτάπητο για να έχουμε συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα. Είπατε κάποιοι από εσά ότι χρειαζόμαστε αποτελέσματα και βεβαίως η υλοποίηση της στρατηγικής μας είναι το κλειδί. Μετά την ε, εξέταση των ε, εκθέσεων στο Συμβούλιο, ε, εξετάζουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο μέχρι την προθεσμία της υλοποίησης των κανόνων της κοινή αγοράς και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα αξιοποιήσουν στο έπακρον αυτό το χρονικό διάστημα για ε, να μην χάσουμε αυτή την προθεσμία. Και σίγουρα και η συζήτηση η σημερινή ήταν πολύ χρήσιμη. Γι' αυτό είναι το λόγο ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό. Τώρα ο συνάδελφος Μπούτζικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, σας ευχαριστώ για όλα σας τα σχόλια. Θα κάνω κάποιες ε, καταληκτικές παρατηρήσεις. Ενώ συζητήθηκε και μάλιστα δύο φορές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ε, το 2011 μέχρι το 2013, υπάρχει υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των Πρωθυπουργών να θέσουν τέλος στην παρουσία των ενεργειακών εισίδων στην Ήπειρό μέχρι το 2015 δηλαδή πρέπει να είμαστε πλήρως διασυνδεδεμένοι. 2015, όχι αργότερα. Πρέπει να έχουμε εξαίρετες διασυνοριακές διασυνδέσεις. Και ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι το εξή. Μία αγορά φιλική προς το χρήστη είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Γιατί θα πρέπει τα πάντα να εστιάζουν στους ε, καταναλωτές μας, είτε τους ιδιώτες, είτε τις εταιρείες, τους εμπορικούς καταναλωτές και όλες οι δυνατότητες με την ε, συνεργασία της βιομηχανίας, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Χρειαζόμαστε νέες λύσεις γιατί Κανένας δεν θέλει να χάνει χρόνο για να ελέγχει τα πάντα στην αγορά. Χρειαζόμαστε και ένα είδος home broker ή distance broker, ενός τέτοιου διαμεσολαβητή, ενός συμβούλου για το πώς ε, θα επιλεγεί ο παραγωγός ή ο διανομέας της ενέργειας. Υπήρχε μια ερώτηση για μια πιο συνεκτική προσέγγιση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την εξόριξη σχιστολιθικού αερίου μπορούμε να πούμε ότι το άρθρο 194 της Συνθήκης της Λισαβόνας δηλώνει ότι κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το δικό του ενεργειακό μείγμα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Φυσικά είναι προφανές. Πρόκειται για την παράγραφο 190. Όμως, σε αυτή τη βάση μπορούμε να πούμε ότι αν ε, υπάρχει διαθέσιμο το σχεστολιφικό αέριο στην Ευρώπη, ίσως πρέπει να προσπαθήσουμε, γιατί θα μπορούσε να βοηθήσει τον ενεργειακό μας κλάδο, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας στο μέλλον. Υπήρχε και μια ερώτηση για τα δίκτυα διανομής και διαμετακόμισης. Θεωρητικά δεν έχει σημασία αν ε, είναι ιδιωτικά ή δημόσια αν ε, το κράτος είναι ο ιδιοκτήτης δηλαδή, γιατί έχουμε ουσιαστικά εδώ την, ε, το unbundling, ε, δηλαδή την αποσύνδεση και θα πρέπει να έχουμε το διαχωρισμό, θα έπρεπε να έχουμε ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση για όλους για όλες τις εταιρείε και από όλες τις χώρες ε, και φυσικά ο μηχανισμός αποζημίωσης εθνικής ε, χωρητικότητας, ικανότητας θα πρέπει να λάβει υπόψη την ενιαία μας αγορά ενέργειας, την κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τι θα κάνουμε με το μηχανισμό αυτό τώρα, πριν ανοίξει πλήρως η αγορά μας. Και Πρόεδρε, δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Ακούσαμε μια σημαντική παρατηρήση από τον κύριο Γκέμπελς για τις ενεργειακές τιμές. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ε, η τιμολόγηση για τις ενεργειακές τιμές και στις επόμενες διαπραγματεύσεις πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Γιατί έχουμε και τις ε, λιανικές αγορές. Πρέπει να δούμε λοιπόν το θέμα της τιμαριθμικής εμπροσαρμογής και χαίρομαι που άκουσα κάποιες παρατηρήσεις από τους συναδέλφους από την Τουρκία και το Κωσυφοπαίδιο για την ενεργειακή κοινότητα. Θέλαμε, θα θέλουμε η Τουρκία όχι να είναι απλώς παρατηρητή στην ενεργειακή κοινότητα, αλλά ως μέλος και είναι σημαντικό να προετοιμάσουμε τη στρατηγική για τα επόμενα δεκαέτη για την ενεργειακή κοινότητα. Και εγώ προσωπικά αισθάνομαι υπεύθυνο και γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Μπούζεκ. Τώρα ο Φιλιπλό, Γενικό Διευθυντή Ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Γκέμπελ θέλει να προσθέσει κάτι, παρακαλώ. Yes, simply... Ναι, ένα ερώτημα και μόνο. Πού είναι η ελεύθερη αγορά όταν έχουμε να κάνουμε με καρτέλ όπως ο ΟΠΕΚ ή όπως ή όπως η γκασπρομ Είναι μακρύς ο κατάλογος. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Φιλιπλό για να απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω είχαμε 22 παρεμβάσεις και μία τώρα 23. Έχω πολλά ερωτήματα. Έχω ξεχάσει ποιο έχει θέσει το καθένα. Με συγχωρείτε. Το πρώτο που θα ήθελα να πω για όλες τις παρεμβάσεις είναι ότι όλοι θέλουμε να επιτύχουμε τους κοινού μας στόχους ε, και να υποφεληθούμε από την ε, ολοκλήρωση της αγοράς ε, στις χώρες μας, όμως λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις επιλογές που κάνουμε επί του ενεργειακού μείγματος, καθώς και το κατά πόσο υπάρχει πραγματική πρόκληση για τη διασύνδεση. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτό ξεκολουθεί να ισχύει ιδίω στην Ανατολική Ευρώπη. Και αυτό καθορίζει και τον αριθμό των ανταγωνιστών στην αγορά. Δεύτερον, αν προσπαθείτε να διαμορφώσετε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να περιορίσετε ε, τις τιμές χρειαζόμαστε μια ανοιχτή αγορά για να έχουμε και ευρωπαϊκούς και μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές και δεν πρέπει να υποτιμούμε τις ε, δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης ε, γηγενών πόρων, ορυκτών καυσίμων όπου υπάρχουν και όπου μπορούν να τύχουν βιώσιμες εκμετάλλευσεις στις ακτές της Βουλγαρίας, ε, στη Ρουμανία, στην Κύπρο. Έχουμε πηγές ε, σημαντικού φυσικού αερίου που πρέπει να αξιοποιήσουμε κατά τη γνώμη μας για να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών που, που είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο. Το δεύτερο, και βεβαίως ε, και για το σχιστολιθικό αέριο, εάν και εφόσον υπάρχει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, εμείς έχουμε εκπονήσει εξολόγηση δεκτύπου και ελπίζουμε τον Ιανουάριο να δημοσιεύσουμε και ανακοίνωση για την εκμετάλλευση του συστολιθικού αερίου. Θα μπορούσε και αυτό να συμβάλλει σε ένα βαθμό αρκεί να θέσουμε τα απαραίτητα κριτήρια βεσιμότητα. Τρίτο στοιχείο για τι ανανεώσιμε. Η ΑΠΕ, όπως ε, αναφέρεται και στον ενεργειακό δικό χάρτη πριν από δύο χρόνια σχεδόν, Όπως και να έχει, υπό οποιοδήποτε σενάριο, θα είναι το βασικό συστατικό ε, της ε, παροχής του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, εάν έχουμε πάρει στα σοβαρά την ε, μείωση ε, της, του διοξιδίου του άνθρακα. γιατί χρειαζόμαστε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας μαζί και με τις ε, πολιτικές ε, ενεργειακής απόδοσης που επίσης είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Αν θέλουμε να έχουμε τις ανανεώσιμες στο σύστημα θα πρέπει να είναι ε, ανταγωνιστικές χωρίς τις επιδοτήσεις όπως και το φυσικό αέριο. Το ίδιο ισχύει όπως και η πυρηνική ενέργεια. Χωρίς επιδοτήσεις θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική για να λειτουργήσει η αγορά. το κύριο στοιχείο και συμπλήρωμα της στρατηγικής δεν είναι μόνο η δημιουργία της ε, ανοιχτής και ελεύθερης αγοράς, αλλά να υπάρχει και ένα είδος ε, αστυνόμευσης, ούτως ώστε οι πηγές ενέργειας να διατίθενται σε ανταγωνιστική βάση. Ανανεώσιμες πηγές χωρίς επιδοτήσεις, ε, εκεί που δεν υπάρχει, εκεί που υπάρχει οριμότητα στην τεχνολογία, να ανοίξουμε την αγορά για τους χώρους όπου δεν υπάρχει ε, οριμότητα, ε, ε, ανάπτυξη της αιωλικής ενέργειας σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, τέτοιες χώρες που έχουν πολύ άνεμο και ήλιο βεβαίως. Και αυτή θα είναι σημαντική συμβολή. γιατί επενδύουμε τόσο πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε χώρες όπου δεν υπάρχουν κατάλληλες καιρικέ συνθήκες είτε στην πλευρά της ε, παροχής, είτε στην πλευρά προσφοράς, είτε στην πλευρά της ζήτησης. Λοιπόν, μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλού άνθρακα. Βεβαίω υπάρχουν δυνατότητε διαφοροποίηση των ε, πηγών ε, προσφορά και αυτό είναι πολύ θετικό. Η διασύνδεση είναι κρίσιμη σημασία και οι μηχανισμοί ικανοτήτων, όπω ανέφεραν αρκετοί, ήταν πράγματι κατακαιρμάτισαν την αγορά εκτός και αν είναι ανοιχτή ε, στις ε, εθνικές ε, πραγματικότητες. Πρέπει πρώτον λοιπόν να καθορίσουμε αν υπάρχει πρόβλημα με τις ικανότητες πριν αναπτύξουμε μηχανισμούς. Κάποιοι είπαν ότι χρειάζεται εναρμόνιση του συστήματος ειδοτήσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρειαζόμαστε περισσότερη πειθαρχία για τους μηχανισμούς ικανοτήτων. Από την Επιτροπή το Νοέμβριο λάβατε κατευθύνσεις και για τα δύο αυτά στοιχεία τα οικονομικά αποδοτικά συστήματα στήριξης και την εισαγωγή των, ε, ικανοτήτων, ε, των μηχανισμών ικανοτήτων. Η Επιτροπή προετοιμάζει κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις το επόμενο καλοκαίρι και πραγματικά ε, μπορεί να επικρίνουμε και τις, τα κράτη-μέλη για τη συμπεριφορά τους, όπως έχουμε κάνει και με τις αντίστοιχες ε, πρακτικές μας για την καταπολέμηση των τραστ. Και πρέπει να εξετάσουμε πότε οι στρεβλώσεις της αγοράς φεύγουν και τους αποτρέπουμε από το να ανοιχτούν στην αγορά. Και τέλος να πω ότι συμφωνώ πολύ με τον πρόεδρο Μπούσεκ, δεν υπάρχει τίποτα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ιδιοκτησία του δικτύου. Βεβαίω το θέμα είναι αν όλοι δρούν δίκαια στην αγορά. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο για την υλοποίηση των κανόνων ανταγωνισμού. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε με τον ΟΠΕΚ και αν μπορούμε να τον ε, συγκρατήσουμε αν θέλετε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό αν είχαμε τα απαραίτητα στοιχεία. Εσείς γνωρίζετε πώς έχει το οικονομικό ε, και πολιτικό στερέωμα. Όμως η Επιτροπή δεν δίστασε να ξεκινήσει ε, εξετάσεις, έρευνες για την προσφορά φυσικού αερίου στην Ανατολική Ευρώπη και μάλιστα και στα δικαστήρια εναντίον βασικών φορέων της αγοράς που δρούσαν στην ε, αγορά ενέργειας στην Ευρώπη με αθέμητο τρόπο που έδρασε ενάντια στον περιορισμό των τιμών. Δεν έχω βρει ακόμα ποιος έγραψε ακριβώς ότι ε, οι τιμές αγοράς της ενέργειας θα πέσουν εξαιτίας ολοκλήρωσης αγοράς. Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία. Ε, Βεβαίω συμφωνώ μαζί σα ότι είναι ανόητο να πει κάποιος κάτι τέτοιο. όμως... Ε, οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί μόνο κατά το ίμιση σε σχέση με άλλες περιοχές. Όλα αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και στην ε, ανακοίνωση για την εσωτερική αγορά ενέργειας, αλλά και στην ανακοίνωση που θα δημοσιεύσουμε στις αρχές του επόμενου έτους. Πολλά μένουν ακόμα να γίνουν, συμφωνώ. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις ε, αγορές λιανικής και πολλοί παρεμβαίνοντες τόνισαν την ανάγκη να ανοίξουν τα συστήματα διανομής και να επικεντρωθούμε σε αποκεντρωμένες μορφές ενέργειας. Αυτό θα βοηθήσει μόνο να ε, μπουν νέοι παίχτες στην αγορά. Πολλά έχουν γίνει. Το γεγονός ότι δεν έχουμε επιτύχει όλους μας τους στόχους δεν σημαίνει πρέπει να τα παρατήσουμε κιόλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ μας ε, έχει μείνει και λίγος χρόνος, καθώς ο Υπουργός ήταν πολύ σύντομος και ο κύριος Μπούζεκ θα ξαναπάρει το λόγο. Ε, ε, ευχαριστώ. Ο συνάδελφός μου Γκέμπελς μας έθεσε σημαντικά ερωτήματα. Συμφωνώ με τα, μαζί σας ότι ε, δεν είναι το θέμα ownership στην ε, νομοθεσία μας. Η ownership όμως το unbundling είναι σημαντική, δηλαδή στο διαχωρισμό της παραγωγής από τα δίκτυα. Και αυτό είναι σημαντικό μια στιγμή όμως πρέπει να εξετάσετε και τις εθνικές περιστάσεις. Εκεί η νομοθεσία προσφέρει ευελιξία, όπως ζήτησε ο αυστριακός φίλος μας, στην εφαρμογή των κανόνων του unbundling. Διαφορετικά συστήματα για τις διάφορες χώρες και μπορούν όντως να οδηγήσουν σε πολύ ε, μεγάλη γραφειοκρατία αν παρασπρώξετε την ownership unbundling. ευχαριστώ, αλλά χωρίς αυτήν δεν, μπορεί να, δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτή ελεύθερη αγορά με ανταγωνισμό. Είναι κρίσιμο θέμα. Θα πρέπει όμως να πάψουμε να ανεχόμαστε τα μονοπόλια στις ε, χώρες μας. Γνωρίζουμε τις χώρες ΟΠΕΚ βεβαίως. Αλλά η Shell Oil στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπτωση δηλαδή αυτή, μπορεί να βοηθήσει λίγο. Και από την άλλη μεριά, αν δείτε τα τελευταία 10-20 χρόνια, παρατηρήσαμε μεγάλες διαφορές στις τιμές του πετρελαίου στις αγορές μας. Ακόμα και με τέτοια ισχυρά μονοπόλια. Να προσθέσω το εξής. Για να αποδυναμώσουμε τα μονοπόλια αυτά από τις καστρόλ χρειαζόμαστε περισσότεροι προμήθεια ενέργειας, περισσότερο αέριο σχιστολιθικό που θα διευκολύνουν να σπάσουν τα μονοπόλια. Να προχωρήσουμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, εγώ δεν έχω άλλη πρόταση για την ώρα. Ευχαριστώ. Ακούσατε και τη διαλεκτική μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Μας έλειπε εδώ το Συμβούλιο και θα κάνουμε τριμερή διάλογο. Γιατί ο συνάδελφος που εκπροσωπεί το Συμβούλιο δεν πήρε θέση. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση για τη συνεισφορά τους. Ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουμε και τις φωνές των Εθνικών Κοινοβουλίων και επίσης να ακούσουν και συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια τις θέσεις του Κοινοβουλίου της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Όπως γνωρίζετε θα συνεχιστεί η συζήτηση στην ίδια αίθουσα σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε στις 3. Και θα προεδρεύσει ο συνάδελφος, ο κύριος Ομετάιτης, και θα συζητηθεί το θέμα της ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη για μια ανταγωνιστική και υφόρο ανάπτυξη. Όλοι οι συγητές που κατέθεσαν την άποψή τους εδώ και όλοι οι συνάδελφοι από τα κοινοβούλια, το επεγραμμίζω αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε προσωπικό. Όλοι λοιπόν οι συνάδελφοι από τα κοινοβούλια καλούνται για το γεύμα στο εστιατόριο των μελών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Αλτιέρο Σπινέλη σε ένα τέταρτο. και το προσωπικό μπορεί να βρει κάποιες άλλες εναλλακτικέ λύσεις στα θεώρια που βρίσκονται τριγύρω. Και καθώς εγώ δεν θα μπορέσω να περιβρεθώ εδώ σήμερα το απόγευμα, θα με αντικαταστήσει ο συνάδελφος. Επομένως, θα ήθελα να σας χαιρετήσω εγώ εδώ είστε στο επανειδήν.